Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα παρακαλώ να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Καλώς ήρθατε και να περάσουμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, την έγκρισή της. Την, είχαμε συμφων... την, σας την είχαμε στείλει 12 Απριλίου και αν δεν υποβληθούν παρατηρήσει ή θεωρούμε ότι εγκρίνεται όπως έχει προταθεί. Περνάμε στο σημείο 2. Να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις και τις επισκέψεις των τελευταίων εβδομάδων. Όσοι ήσασταν στην επίσκεψη στην Αθήνα, ίσως ε, ζητήσουν το λόγο, αλλά ας αφήσουμε τη συζήτηση για την Αθήνα αργότερα, όταν θα εγκρίνουμε την έκθεση στην Επιτροπή. Εγώ απλώς να σας πω εν συντομία ότι μία αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας μετέβη στην Αθήνα την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν το ΕΛ και οι σοσιαλιστές και δημοκράτες, οι φιλελεύθεροι και οι ΓΚΟΕ. Αυτές οι ομάδες έστειλαν εκπροσώπους στην αντιπροσωπεία της ΑΦΚΟ στην Αθήνα. Είχαμε πολύ καρποφόρες ε, και επικοδομητικές ε, συναντήσεις και ανταλλαγή απόψεων με δύο μόνιμες επιτροπές ε, της Βουλής των Ελλήνων, την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Επίσης, είχαμε συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, με τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων και τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικράτειας είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο και είναι και με, μερικές φορές αντίστοιχο και με συνταγματικό δικαστήριο σε κάποιες χώρες. Επίσης συζητήσαμε και με πολλούς εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας πανεπιστημιακούς. Πολύ χρήσιμη επίσκεψη, όχι μόνο γιατί ενημερωθήκαμε για τις ε, ανησυχίες της Ελλάδας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή και μάλιστα πριν την ε, συνάντηση με τους εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση του προγράμματος, οπότε υπήρχε έντονο ενδιαφέρον και για θέματα που μας αφορούν, δηλαδή τις σχέσεις εθνικών αρχών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και το θέμα της συνταγματική νομιμότητας, της συνταγματικότητας δηλαδή των εθνικών μέτρων. Μάλιστα, ακούσαμε πολλά σχόλια από τους Έλληνες ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Συμφωνήσαμε ιδιαίτερως ε, με τους βουλευτές για την ανάγκη να κρατήσουμε στενές επαφές και μάλιστα προσκαλέσαμε τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες για ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής. Μάλιστα μετά την Αθήνα είχα προσκληθεί και μία διάσκεψη στη Ρώμη στα πλαίσια της διαδικασίας που ξεκίνησε η Βουλή των Αντιπροσώπων και η πρόεδρος της Λάουρα Μπολντρίνη με θέμα το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πολλοί εθνικοί βουλευτές ε, συνυπέγραψαν μαζί με τους Ιταλούς βουλευτές μία διακήρυξη για την ε, ε, πιο ενισχυμένη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ακολουθητέα πορεία. Μάλιστα και στην συνέχεια πολλοί άλλοι εθνικοί βουλευτές συνυπέγραψαν αυτή τη διακήρυξη. Και υπάρχει τέτοια κινητοποίηση από πολλά εθνικά κοινοβούλια. Είχαμε συζητήσεις και με τον Φραν Τίμερμανς, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ολλανδικής Κυβέρνησης, τον κύριο Κούντερς, αλλά και με εκπροσώπους ε, προηγούμενων και επόμενων προεδριών της Σλοβακικής Προεδρίας, τον Αντιπρόεδρο της Μάλτας. Και το μόνο που μπορώ να σας πω μετά τη συζήτηση είναι ότι οι εθνικές κυβερνήσεις βέβαια δεν είναι τόσο προσανατολισμένες προς το μέλλον και με τις θεσμικές αδυναμίες και τις ε, μακροπρόθεσμες ε, προκλήσεις. Περισσότερο είναι προσανατολισμένοι σε κυβερνήσεις το εδώ και τώρα δηλαδή στο βραχυπρόθεσμα πώς θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Πάντως θα συνεχιστούν αυτές οι συζητήσεις Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στο μέλλον. Ε, επίσης, ε, έχουμε επιτέλους ε, την έγκριση της διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάτι που περιμέναμε διακαώς εδώ και πολύ καιρό, τις αλλαγές δηλαδή στους κανόνες για τις ε, εφαρμοστικές εκθέσεις. Επισταμμένως ε, ζητούσαμε, για να μην πω ότι δίναμε μάχη, ήταν πολύ σημαντικό για μας αυτό το θέμα, ώστε τα πιο καθόδη ζητήματα να τα συμπεριλάβουμε στο πεδίο εφαρμογής των εκθέσεων ε, εφαρμογής, γιατί κάτι τέτοιο δεν ίσχυε γιατί αυτή ήταν η βασική, αυτή ήταν η βασική μας στόχη. Ε, γιατί μέχρι τώρα μόνο η εφαρμογή ευρωπαϊκού δικαίου από τα κράτη-μέλη θεωρούνταν ότι επιτροπόταν σε αυτές τις εφαρμοστικές εκθέσεις. Τώρα έγινε κάποια διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή τους. Ζητήσαμε μάλιστα και άδεια και έχουμε πια την αξιοδότηση και μπορούμε να εκπονήσουμε τις πρώτες δύο τέτοιες εφαρμοστικές εκθέσεις Ήδη από πέρυσι τον Οκτώβριο είχαμε ζητήσει τη σχετική εξουσιοδότηση. Η πρώτη τέτοια έκθεση εφαρμογής αφορά την εφαρμογή των διατάξεων των συνθηκών για τα Εθνικά Κοινοβούλια και τον Οκτώβριο αναθέσαμε την έκθεση αυτή στον Πάολο Ρανζέλ και η δεύτερη εφαρμοστική έκθεση αφορά την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο. Την έκθεση τη διεκδίκησε η Γκούε και η συγγήτρια είναι η κυρία Μπάρμπαρα Σπινέλη. Οπότε επιτέλους μπορούν οι δύο να ξεκινήσουν το έργο τους. Υπάρχει ανοιχτό και το θέμα της ενεργούς συμμετοχής μας στην εκπόνηση της εφαρμοστικής έκθεσης για την εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας. Η Γραμματεία μάλιστα θα σας στείλει τους νέους κανόνες για τις εκθέσεις αυτές, ε, τις εκτελεστικές, οι εφαρμοστικές και οι συντονιστές ε, θα ασχοληθούν πιο συγκεκριμένα για τα θέματα αυτά. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης, της 14ης Ιανουαρίου δηλαδή του 2016. Αν μέχρι το τέλος συνεδρίασης δεν υποβληθούν ενστάσεις ή παρατηρήσεις θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα τα πρακτικά. Και περνάμε στο κυρίως θέμα της πρωινής μας συνεδρίασης, που είναι η δημόσια ακρόαση με θέμα την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κάποιος απολογισμός μετά τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της ευρωπαικης ενωσης στην ευρωπαικη συμβαση ανθρωπινων δικαιωματων καποιο απολογισμος Ένωσης και θα συζητήσουμε και την ακολουθητή απορία. Έχουμε προσκαλέσει πολλούς εμπειρογνώμονες και να σας πω δύο λόγια για να σας υπενθυμίσω το λόγο της διοργάνωσης αυτής της δημόσιας ακρόασης. Όπως ξέρετε, η, Επιτροπή έχει ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μία γνωμοδότηση με θέμα τη συμβατότητα του σχεδίου συμφωνίας με τα συμβαλώμενα μέρη που είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και ζήτησε από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να αποφανθεί κατά πόσο η, το σχέδιο αυτό της Συμφωνίας Προσχώρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συμβατό με τις συνθήκες. Η γνωμοδότηση του δικαστηρίου ήταν αρνητική. Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων έγινε το Δεκέμβριο του 2014, αμέσως μετά τη δημοσίευση της γνωμοδότησης ακολούθησε ανταλλαγή απόψε με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, με τη νομική μας υπηρεσία, τη νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα έχουμε εκπροσώπους ε, όλων αυτών των υπηρεσιών σήμερα στη δημόσια κρόση. Το, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έκρινε μη συμβατή τη συμφωνία, το σχέδιο συμφωνίας με τις συνθήκες. Έχει περάσει σχεδόν ένα χρόνος από την υιοθέτηση της γνωμοδότησης του ΔΕ και ελπίζουμε ότι υπήρξε κάποια εξέλιξη ε, στις συζητήσεις και στην προσέγγιση. Και θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα τους εμπειρογνώμονές μας, τους καλεσμένους μας. Θα, στους, θα σας παρουσιάσω όταν θα τους δώσω το λόγο. Δυστυχώς ένας από αυτούς ο καθηγητής Ρουι Μανουέλ Μόουρα Ράμος από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κοίμπρα στην Πορτογαλία που ήταν και πρώην δικαστής του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην πρόεδρος του Πορτογαλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου και τον περιμέναμε πώς και πώς στη δημόσια κρόση. Δυστυχώς, λόγω ασθενείας, δεν μπόρεσε να μεταβεί στις Βρυξέλλες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη δημόσια ακρόαση αρχής γενομένης από τις Προεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον εκπρόσωπο της Προεδρίας, στον κύριο Μαρτέιν Ντεχράβε, που είναι επικεφαλής του Τμήματος Νομικών και Θεσμικών Υποθέσεων και συντονιστή δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων στη μόνιμη Ολλανδική Αντιπροσωπή στι Βρυξέλλε. Κύριε Ντεχράβε, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ καταρχήν κυρία Πρόεδρε για την πρόσκληση για συμμετοχή σε αυτή τη δημόσια κρόση για να σα παρουσιάσω τη θέση του Συμβουλίου. Γιατί είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε ένα απολογισμό τη κατάσταση και να δούμε την ακολουθητέα πορεία μετά το χρόνο που πέρασε από την γνωμοδότηση. Η τελευταία μα συνεδρίαση ε, και ανταλλαγή απόψεων είχε λάβει χώρα μετά την ε, δημοσίευση τη γνωμοδότησης του δικαστηρίου 2 13 που ε, χαρακτήρισε το σχέδιο συμφωνίας ε, μη συμβατό με τις συνθήκες. Φυσικά είναι περιττό να σας Όπω ε, απογοητευτήκαμε στο Συμβούλιο, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι συνέπειε όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται. Είναι σαφέ μετά τη γνωμοδότηση ότι υπάρχει ανάγκη έναρξη των διαπραγματεύσεων στο Στρασβούργο. Θα πρέπει όμω να γίνουν και τεχνικέ προεργασίε για να ετοιμαστούμε για τι επόμενε διαπραγματεύσει. Και όπω είπατε, ε, αυτό το εγχείρημα θα είναι χρονοβόρο. Και μετά από μια περίοδο προβληματισμού συνεχίσαμε τις συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο ώστε να βρούμε λύσεις στα τεχνικά ζητήματα που επισήμανε το δικαστήριο και, το Ευρωπαϊκό, ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως διαπραγματευτής ε, είχε διαβουλεύσει με την Ειδική Επιτροπή που όρισε ε, το Συμβούλιο για, την, για τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα δικαιώματα και την ελεύθερη διακίνηση με για να εξεταστεί η γνωμοδότηση. Και κατά την προηγούμενη λεπτονική Προεδρία πολλά ε, τεχνικά, διαδικαστικά, δικονομικά ζητήματα εξετάστηκαν. Για παράδειγμα, ε, το θέμα της, του μηχανισμού παθητικής ομοδικίας, ε, η αλληλέγγυα ευθύνη εναγωμένου και συναναγωμένου η προηγούμενη ε, συμμετοχή, η προηγούμενη εξέταση του δικαστηρίου τα θέματα 3 και 44, το θέμα του πρωτοκόλου 16 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και οι σχέσεις ε, του άρθρου 53 της, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του άρθρου 53 της ΕΣΔΑ, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όλα αυτά τα σημεία επισημάνθηκαν στην κοινομοδότηση του ΔΕΕ, του Δικαστηρίου Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα γίνει θα επιδιώξουμε τεχνική πρόοδο, σημαντική πρόοδο σε αυτά τα τεχνικά θέματα. Βέβαια, εκκρεμούν τα πιο δύσκολα θέματα, τη ΣΚΕΠΑ και τις αμοιβέ εμπιστοσύνη. Και μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει την ανάλυση της για τα θέματα αυτά, με πιθανέ ε, προτάσεις και επιλογές, ε, θα, ε, θα τα εξετάσουμε κατά προτεραιότητα στο Συμβούλιο. Κυρίε και κύριοι, το Συμβούλιο στις 9 Οκτωβρίου του 2015 οι Υπουργοί Δικαιοσύνη διατράνωσαν την δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στη Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπω προβλέπουν οι συνθήκε. Οπότε μπορείτε να υπολογίσετε στην πλήρη δέσμευση του Συμβουλίου ε, για να πραγματοθεί η προσχώρηση. Και με αυτή την άποψη θα ήθελα να βοηθήσω την πρόοδο και τα μέλη τη Επιτροπή για την αμέριστη υποστήριξη που μας δείχνεται και για την οργάνωση αυτής της ε, δημόσιας ακρόσης που θα είναι πολύ χρήσιμη για την ακολουθητέα μας πορεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα δίνω το λόγο στον Χάνες Κρέμερ, τον οποίο έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν και κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων, αλλά και κατά τη διάρκεια της πρώτης ανταλλαγής απόψεων που είχαμε μετά την κοινοποίηση της γνωμοδέωτησης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήσασταν ή είστε ο επικεφαλής διαπραγματευτής. Ήσασταν σε κάθε περίπτωση υπεύθυνο για τις διαπραγματεύσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπροσωπείτε σήμερα τη νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τα θετικά σας λόγια, για την πρόσκλησή σας στη σημερινή συνεδρίαση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητά τα θέματα αυτά και το βλέπουμε σήμερα με την ένταξη του σημείου αυτού στην ημερήσια διάταξη. Ήδη ο κύριος Δεγκράβα περιέγραψε την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα δηλαδή, θα ήθελα εγώ να φωτίσω λίγο την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλωστε εμεί ζητήσαμε τη γνωμοδότηση αυτή από το Δικαστήριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει προσιλωμένη στην προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υφίσταται νομική η υποχρέωση για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνάψουν συμφωνία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βάσει βέβαια των προδιαγραφών και των όρων που προβλέπονται στις συνθήκες και συγκεκριμένα στο πρωτόκολλο 8 της συνθήκης. Η προσχώρηση αυτή θα οδηγήσει σε μια περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των θεμελιδών δικαιωμάτων, θα καταστήσει τον νοσιακό δίκαιο πιο ισχυρό και θα καταστήσει και πιο συνεκτική την προστασία των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η προσχώρηση Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παραμένει ένας πολύ σημαντικός στόχος. Βέβαια, η γνωμοδότηση της 18 Δεκεμβρίου του 2014, του δικαστήριου δηλαδή, θέτει κάποια πολύ σοβαρά νομικά ζητήματα, ορισμένα εκ των οποίων είναι πολύ πολύπλοκα από νομικής και πολιτικής πλευράς θα μπορούσα να φέρω τα δύο σημεία τα οποία ανέφερε και η Προεδρία του Συμβουλίου, συγκεκριμένα την ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια και το ζήτημα της αμοιβέ εμπιστοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο χρειάστηκε να περάσει μια περίοδος περισυλλογής προκειμένου να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος από νομικής και πολιτικής πλευράς για να προχωρήσουμε το ζήτημα αυτό. Επί του παρόντος και μετά την ολοκλήρωση της Τετωνική Προεδρίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ως επίσημος διαπραγματευτή ε, για το ζήτημα αυτό συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με την Ειδική Επιτροπή του Συμβουλίου για τα διάφορα ζητήματα, τα εκρεμή ζητήματα, τα οποία μπορούμε να δούμε στη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελευταία σχετική συνεδρίαση έγινε στις 4 Νοεμβρίου 2015 και η επόμενη συνεδρίαση προβλέπεται την επόμενη εβδομάδα στις 26 Απριλίου συγκεκριμένα. Επί του παρόντος, όπως ήδη είπε ο πρόσωπος της Προεδρίας, οι διαβουλεύσεις αυτές επικεντρώνονται στα πιο τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα. Η Προεδρία ήδη απαρίθμησε όλα αυτά τα ζητήματα. Σε ένα μεταγενέστερο βέβαια στάδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις, πιθανούς τρόπους δηλαδή, στα πλαίσια της διαβούλευσης για να επιληθούν ζητήματα όπως η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και το ζήτημα της αμοιβέ εμπιστοσύνη. Στόχος του όλου εγχειρήματο είναι να καταφέρουμε να δούμε ποια θα είναι η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις ε, τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν στο σχέδιο συμφωνίας προσχώρησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου του Ιουνίου του 2010 προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τα συμβαλόμενα μέρη στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Και εφόσον μιλάμε για το άνοιγμα εκ νέου των διαπραγματεύσεων, πρέπει να σα πω ότι οποιασδήποτε τροποποιήσει στο σχέδιο συμφωνία προσχώρηση που θα ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περιορίζονται πολύ αυστηρά στο απολύτω αναγκαίο προκειμένου να ικανοποιηθούν οι περαιτέρω απαιτήσει οι οποίε προβλήθηκαν μέσω τη γνωμοδότηση 2.13 του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μελλοντικέ λοιπόν διαπραγματεύσει για τι απαιτούμενε αυτέ τροποποιήσει θα λάβουν χώρα σε πλήρη διαβούλευση με την Ειδική Επιτροπή του Συμβουλίου και βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πλήρως ενημερωμένο για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Και πρέπει να πω ότι στηριζόμαστε και στη δική σας τη συμβολή και την υποστήριξη, που από πολιτικής πλευράς είναι πάρα πολύ σημαντική. Γνωρίζουμε ότι είστε στο πλευρό μας, ότι είστε ένα σημαντικό σύμμαχος των υπολείπων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ας περάσουμε τώρα στην άλλη πλευρά, αν θέλετε. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η άλλη πλευρά στην όλη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, σε απευθυνθούμε τώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ας πούμε, το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι η άλλη πλευρά, η απέναντι όχθη. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο Πολάκης Κίφς, ο οποίος ε, είναι σύμβουλος, νομικός σύμβουλος για τα νομικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Δεν ξέρω αν ε, Πραγματικά είναι αυτός, αυτή η θέση σας η οποία βλέπω εδώ πέρα στην ημερήσια διάταξη. Είστε διευθυντή και υπεύθυνο για ζητήματα νομική φύση στα πλαίσια του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα εδώ σήμερα. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Όπω αναφέρθηκε ευθύ εξ αρχή, θα σα προσφωνήσω ω νομικό σύμβουλο του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Πρέπει να τονίσω όμω ότι σε σχέση με αυτή την τοποθέτηση, τοποθέτηση α, όσον αφορά την γνωμοδότηση υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την επίσημη αυτή ε, εκπροσώπηση κάνοντας λόγο για την ε, ε, γνωμοδότηση αναμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις πώς μπορούν οι διάφορες ενστάσεις ε, να ε, ξεπεραστούν. Είμαστε ευγνώμονες στην Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή που μας προσκαλέσατε να συμμετάσχουμε σε αυτή την συνεδρίαση. Σίγουρα δεν είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης που θα πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα ξεπεράσει τα εσωτερικά της προβλήματα. Οπωσδήποτε, οποιαδήποτε πρόταση και να υποβληθεί θα αποτελέσει αντικείμενο προφανώς διαπραγματεύσεων στο Στρασβούργο και σε σχέση με τα όσα έχουν γίνει από πλευράς και αναφέρθηκαν από τον κύριο Hans Κρέμερ συνάδελφό μου και από πλευράς των θεμάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μια και τα θέματα είναι πολύ άριθμα και σύνθετα ε, υπάρχει και η ε, γραπτή έντυπη παρέμβαση. Τώρα θα επικεντρωθώ σε κάποια από αυτά τα ζητήματα. Η Γενική μου Συμβουλή, αν μου ζητούσατε ως νομικού συμβούλου τη Συμβουλή μου, μπορεί να συμπεριληφθεί στα εξή πέντε σημεία. Πρώτον, να υπάρξουν ε, περιορισμοί όσον αφορά τις τροποποιήσεις για την προσχώρηση διότι ο πραγματικός κίνδυνος όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα για τις αρμοδιότητες του, του ε, Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με αυτόν τον τρόπο θα περιόριζε τις δραστηριότητες και θα υπονόμευε τις ε, δραστηριότητες του. Δεύτερον, μην χρησιμοποιήσετε θέματα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν ε, αντικείμενο περιπλοκής Τρίτον, να αποφευθούν διατάξεις για τις εσωτερικές διεργασίες όσον αφορά διεθνείς συμβάσεις ε, στα οποία, στις οποίες ε, τα, ε, μπορεί να υπάρχει ζήτημα από πλευράς των κρατών μελών. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εσωτερικοί κανόνες και κανονισμοί ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να συμμορφώνονται με το κοινοτικό δίκαιο. Και τελευταίο και πέμπτο σημείο, οι ερμηνευτικές δηλώσεις εφόσον δεν μπορούν να αποφευθούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο. Η συνθήκη, σύμβαση προσχώρησης μπορούν να δώσουν, μπορεί να δώσει δικαιώματα και στο πρωτογενές και στο δευτερογενές δίκαιο να δράσουν. Ε, σε κάποια συγκεκριμένα θέματα όσον αφορά το πρωτόκολλο 16 και τη διάταξη των, για τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τέτοια θέματα προς ε, διευθέτηση στο, στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Αυτά τα θέματα είτε μέσω μονομερών δηλώσεων είτε μέσω ε, προσαρμογών μια και η, ε, τα πλαίσια του το πρωτοκόλλου 16 δεν είναι δεσμευτικά πρέπει να πούμε ότι είναι ήδη σημαντικό ότι τρία κράτη-μέλη έχουν ήδη προ, ε, επικυρώσει το πρωτόκολλο 13 χωρίς οποιασδήποτε ερμηνευτικές δηλώσεις για να μπορέσει η δήλωση όσον αφορά τις ε, εσωτερικές ε, τριβές ε, να μπορέσει να λειτουργήσει θα πρέπει ο ευδιάκτητος ρόλος όσον αφορά την ερμηνεία του δικαίου να μπορέσει να λειτουργήσει με θετικό τρόπο η ένσταση όσον αφορά την συμμόρφωση του άρθρου 53 και με την χάρτα ήταν μια έκπληξη και για όσους γνωρίζουν τα θέματα του δικαίου πώς μπορεί μια τέτοια σύμβαση να αναγεννήσει, να αναζωογονήσει δικαιώματα τα οποία έχουν απεμποληθεί ήδη από τα κράτη-μέλη. Το άρθρο 53 επιτρέπει σε συμβαλόμενα κράτη-μέλη να διασφαλίζουν το ανώτατο επίπεδο προστασίας. Αυτή η διάταξη δεν αφορά αρμοδιότητες ή εξουσίες είναι απλά και μόνο ένας κανόνας που δίνει την δυνατότητα να είμαστε πιο λειτουργικοί μέσα στο πλαίσιο αυτό. Όσον αφορά την αμοιβαία εμπιστοσύνη, αμοιβή εμπιστοσύνη βασιζόμαστε σε αυτές τις αρχές και αξίες. Ο σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα είναι κέριο σημείο για ε, το δίκαιο και τα κράτη-μέλη έχουν ε, οποιασδήποτε ε, διαπιστώσεις ε, γίνονται για τέτοιες παραβιάσεις πρέπει να δρούν. Έχουμε και τις προδιαγραφές που εφαρμόζονται σε αυτό το πεδίο. Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας κατέληξε σε μια απόφαση την 15η Δεκεμβρίου 2015 το ίδιο ακριβώς συμπέρασμα στο οποίο είχε καταλήξει το δικαστήριο του Στρασβούργου, δηλαδή ότι οι εθνικές αρχές έχουν το καθήκον ώστε σε κάποια ατομική περίπτωση να διασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα των ατόμων θα είναι σεβαστά ε, Καλωσορίζουμε αυτή την απόφαση αναγνωρίζοντας ότι η εκτέλεση θα πρέπει εδώ οπωσδήποτε όσον αφορά μια ταπεινωτική μεταχείριση να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Η ένσταση θα μπορέσει αντίστοιχα με αναπερίπτωση να ε, συμπληρωθεί και με διάλογο μεταξύ ε, του δικαστηρίου και των ε, αρμοδίων όταν αυτό θα είναι αναγκαίο να υπάρξουν συγκεκριμένες διατάξεις για την αναγνώριση αυτών των περιπτώσεων. Επόμενο σημείο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια ολόκληρη σειρά συγκεκριμένων προτάσεων πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τέτοιου είδους ενστάσεις και επιφυλάξεις. Δεν θα ήταν εύθετο για μένα να σχολιάσω αυτές τις περιπτώσεις χωρίς να μου ζητηθεί να το πράξω. Θέλω να υπενθυμίσω ότι οι αντίστοιχες αυτές διατάξεις είχαν συνταχθεί ώστε να μπορέσει να διασφαλίζεται η αυτονομία της, Ευρω... της ε, ε, ευρωπαϊκής νομικής τάξεως πραγμάτων ώστε να μην υπάρχει μονομερής επέμβαση από πλευράς του όταν ε, θέλουμε να προχωρήσουμε δεν πρέπει να θυσιάζουμε τις αρχές ε, που μας διέπουν. Και τέλος η τελευταία ένσταση όσον αφορά την ΚΕΠΑ αυτή η ένσταση αφορά ακριβώς τον πυρήνα του συμβιβασμού στον οποίο καταλήξαμε για την ε, Συμφωνία Προσχώρησης. Το να υπάρξει μια εξαίρεση δεν μπορεί να συνάδει με την ιδέα μιας ε, ευρείας ε, λειτουργίας αυτής της χάρτας και αυτής της σύμβασης. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει αυτό να το λάβουμε απόλυτα υπόψη. Μια πιθανή λύση θα μπορούσε να ήταν μια δήλωση στην διακυβερνητική διάσκεψη ώστε να μπορέσει έτσι να διατυπωθεί η προσχώρηση ώστε το δικαστήριο να μπορεί να επιλαμβάνεται όλων των υποθέσεων ε, που το αφορούν από πλευράς μας. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με βάση την δήλωση του Προέδρου Γιούγκερ όσον αφορά την προσχώρηση που είναι καθήκον και προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλωσορίζουμε ιδιαίτερα και την δήλωση που έγινε από πλευράς του κυρίου Κρέμερ, του συναδέλφου το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σίγουρα δεν διευκόλυνε το έργο μας ε, όχι μόνο λόγω της εμβέλειας αλλά και λόγω των θεμάτων της, ε, των νομικών επιπτώσεων. Ένας πρώην δικαστής ε, του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περιέγραψε την απόφαση αυτή ως μια πολιτική απόφαση που περιγράφει νομικά ζητήματα. Και γι' αυτό όχι μόνο σε σχέση με την ε, προσχώρηση αλλά και με την ίδια τη συνθήκη θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις ε, ε, τροπολογίες. Αυτό μπορεί να είναι μια επίλυση αλλά υπάρχουν και αμφιβολίες, ισχυρές αμφιβολίες. Όπου είναι δυνατόν θα πρέπει με ρεαλιστικό τρόπο να αντιμετωπίζονται οι ενστάσεις αναμία εκάστοτε ταυτοποιώντας τις λύσεις που θα σέβονται και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και την ε, ακαιρεότητα του ε, συστήματος λειτουργίας ε, του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η ολοκλήρωση μιας αναθεωρημένης διατύπωσης μέσων θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε οι λύσεις να μπορούν να και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Θα κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε να προχωρήσει αυτό το θέμα, αναφέρθηκε. Η δική μου παρουσία είναι ένα ενθαρρυντικό, προτρεπτικό μήνυμα. Α συνεργαστούμε για να επιτύχουμε το κοινό, κοινό μας στόχο. Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη, υπέρ των πολιτών τη Ευρώπη. Σα ευχαριστώ. Um, uh, ευχαριστώ πολύ πολύ, αγαπητέ κύριε Πολακέβιτς. Μία ακόμη πληροφορία που ξέχασα να την κάνω στην αρχή. Καλέσαμε και τον κύριο Κεν Λέναρτς, τον πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για προφανείς λόγους ε, δεν ήρθε. Το δικαστήριο κρίνει ότι δεν είναι σκόπιμο να σχολιάζει τις συνέπειες των ίδιων του το γνωμοδοτήσεων. Εύλογο και το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε. Και όταν είπατε κύριε Διευθυντά ε, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί θα έλεγα, ό,τι απαιτείται. Αυτό εννοούσε ο κ. Γιάκμεν, ότι θα κάνει ό,τι μπορεί, δεν θα αφιστεί προσπαθειών. Και το εκτιμούμε ιδιαίτερος. Περνάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Ζαν Πολ Ζακέ, που είναι επίτιμος Γενικό Διευθυντής τη Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου. Με μακρά πανεπιστημιακή σταδιοδρομία και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, ε, στο οποίο διατέλεσε πρόεδρος και ε, ήταν και πρόεδρος στο Κολέγιο τη Ευρώπη. Κύριε Ζακέ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σα ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Θα ήθελα τώρα να κάνω σύντομα δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την ΕΣΔΑ. Κατά τη γνώμη μου, η μη προσχώρηση είναι χειρότερη από αυτά που αναγγέλει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΔΕΕ. Γιατί όλες οι ενστάσεις ε, ε, που υπέβαλε το Δικαστήριο κατά της προσχώρησης θα γυρίσουν μπούμεραγκ κατά τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά των κρατών μελών σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η προσχώρηση. Και θα σας κάνω μια ε, σύντομη περιγραφή. Το δικαστήριο είπε ότι η συμφωνία δεν σεβόταν την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Στην παρούσα όμω κατάσταση σήμερα τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Το ΕΔΑ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι απόλυτος ε, κύριος και δικαστής να κρίνει τι εμπίπτει στις ε, κοινωτικές αρμοδιότητες και στην ε, νομολογία του από μια υπόθεση φωσφορίου. ήταν ε, σαφώς κυρίαρχο να αποφασίσει τι είναι και τι όχι στις κοινοτικέ αρμοδιότητες. Επίσης, το ΔΕ λέει ότι δεν μπορεί το δικαστήριο να αποφαίνεται σε προδικαστικό ζήτημα πριν αποφανθεί αντίστοιχα το ΕΔΑ για το θέμα αυτό. Κάθε μήνα όμως βλέπω αποφάσεις του ΕΔΑ, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που ερμηνεύουν και εφαρμόζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κληθεί για να αποφανθεί στα πλαίσια της προδικαστικής παραπομπής. Επίσης, ε, το ΔΕ, το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας λέει ότι σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των κρατών μελών αυτές ε, θα επιλύονται στο Στρασβούργο αντί να επιλύονται στα πλαίσια των συνθήκων. Αλλά ακόμη και τώρα αυτό είναι δυνατό για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και θα μπορούσα να συνεχίσω με πολλά παραδείγματα ακόμη για να σας αποδείξω ότι οι ενστάσεις του, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάζουν τα κράτη-μέλη σε πολύ χειρότερη θέση από αυτή που θα βρίσκονταν αν είχε γίνει δεκτή η συμφωνία ή το σχέδιο συμφωνίας προσχώρησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν θα καταδικαζόταν στο ΕΔΑ, γιατί δεν, ήταν, ε, δεν θα ήταν μέλος της σύμβασης. Τα κράτη-μέλη όμως όταν εφαρμόζουν ε, το ενωσιακό δίκαιο δίνονται να προσεχθούν και να καταδικαστούν από το ΕΔΑ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οπότε με την γνωμοδότησή του το δικαστήριο φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τα κράτη-μέλη και ε, ε, είτε τα αναγκάζει να παραβιάσουν το ενωσιακό δίκαιο για να εφαρμόσουν την ΕΣΔΑ, είτε να παραβιάσουν την ΕΣΔΑ για να εφαρμόσουν το ενωσιακό δίκαιο. Και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητικό. Γιατί ε, για το δημοψήφισμα στο Γιβραλτάρ, το Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε ακριβώς σε αυτή την κατάσταση και η λύση ήταν πολύ δύσκολη. Γι' αυτό είναι επίγον για να διασφαλιστούν τα κρατη και να μπορέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπαχθεί σε έλεγχο, να ξανακαθίσουμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Και σε αυτή την Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων αντιμετωπίζουμε δύο είδη προβλημάτων. Τα εύκολα και τα ιδιαίτερως δυσεπίλητα προβλήματα. Και το εγχείρημα και το διάβημα που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να ξεκινήσει από τα πλούστερα και τα ευκολότερα θέματα και να περιμένει αργότερα να προλιαθεί το έδαφος για τα πιο δυσεπίλητα. Ποια είναι τα απλά θέματα. Όλες οι τεχνικές ενστάσεις του δικαστηρίου, του ΔΕ, που αφορούν ε, το μηχανισμό της ε, συνυπευθυνότητας ή της παθητικής ομοδικίας, την ε, προηγούμενη εξέταση από το δικαστήριο, το άρθρο 33 του ΕΣΔΑ, μάλλον 53 εννοεί ο μιλητής, του ΕΣΔΑ και του χάρτη. Τα θέματα που αφορούν τα κράτη-μέλη και τις συμβουλευτικές γνωμοδοτήσεις που μπορούν να ζητηθούν από το Δικαστήριο του Στρασβούργου. Για όλα αυτά τα θέματα, με μικρές αλλαγές τεχνικές, θα μπορούσαμε να λύσουμε τα προβλήματα και σε μερικές περιπτώσεις, ακόμη και με ερμηνευτικές δηλώσεις θα μπορούσαμε να λύσουμε αυτές τις ενστάσεις. Δύο είναι τα πιο δυσεπίλητα, τα πραγματικά δυσεπίλητα ζητήματα. Το πρώτο αφορά την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και γιατί είναι δυσεπίλητο. Γιατί το θέμα της αμοιβαία εμπιστοσύνη δεν συνδέεται με τη συμφωνία προσχώρησης και μάλιστα είναι και περίεργο που το αναφέρει καν το ΔΕ. Γιατί δεν εμπίπτει στη συμφωνία αφορά τη διαφορά της νομολογίας των δύο δικαστηρίων. Γιατί τα δύο δικαστήρια, το ΕΔΑ και το ΔΕ, δεν ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και δεν ξέρω αν μπορούμε το ζήτημα αυτό να το επιλύσουμε με μια συγκεκριμένη διάταξη, όπως μας είπε ο κύριος Πολακέβιτς, γιατί για τις διαπραγματεύσεις χρειάζονται δύο μέρη. Και μια τέτοια ρητή διατύπωση δύσκολα θα ήταν δεκτή από το ένα μέρος. Και ίσως ε, τα δύο δικαστήρια θα μπορούσαν να συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση. Η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και την Αμοιβαία Εμπιστοσύνη έδειξαν ένα σχετικά δηλό και μετριοπαθές βήμα αντάξιο της εικόνας του ΔΕ. Περιμένουμε απόφαση και του δικαστηρίου του Στρασβούργου για τα ίδια θέματα. Κάθε δικαιοδοτικό όργανο, κάθε δικαιοδοσία μπορεί να κάνει κάποια βήματα για να συγκλίνει τις θέσεις του με αυτές του άλλου δικαιοδοτικού οργάνου. Και απομένει το τελευταίο θέμα, το θέμα της κοινή εξωτερικής πολιτικής και κοινή πολιτικής ασφάλειας. Αυτό όντως είναι δύσκολο. Το να αποκλείσουμε την ΚΕΠΑ, την κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή πολιτική ασφάλειας από το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας κατά τη γνώμη μου είναι απαράδεκτο για τα υπόλοιπα συμβαλόμενα μέρη της σύμβασης, της ΕΣΔΑ. Οπότε τι με έλεγενέστε, τροποποίηση, αναθεώρηση της συνθήκης. Όνειρο απατηλό, βέβαια δεν απαγορεύονται τα όνειρα, αλλά μάλλον απίθανο μου φαίνεται σχετικά σύντομα. Ίσως θα μπορούσαμε να περιμένουμε μία εξέλιξη της νομολογίας, γιατί εκκρεμούν δύο ζητήματα στο δικαστήριο για τις αρμοδιότητες, της, τις αρμοδιότητες τους προς την ΚΕΠΑ και θα δούμε αν εκεί υπάρχει κάποια δυνατότητα ανοίγματο ή όχι. Αλλά για αυτό το σημείο, για την ΚΕΠΑ, είναι που θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Εγώ θεωρώ ότι η λύση που προκρίνει το σχέδιο συμφωνίας ήταν πολύ έξυπνη γιατί προβλέπει ότι και σε θέματα ΚΕΠΑ και σε άλλους τομείς ε, μπορούσαν να προσβληθούν στο δικαστήριο ε, πρώτα τα κράτη-μέλη και ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συμμετέχει ως συναγόμενη μαζί με τα κράτη-μέλη. Οπότε άφηνε στη διακριτική ευχαίρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να κρίνει αν ήθελε η ίδια να περιληφθεί στην παθητική ομοδικία για θέματα ΚΕΠΑ στο δικαστήριο. Ήταν πολύ έξυπνη λοιπόν αυτή η λύση, δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πάντως ότι αν το δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο να κρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ΚΕΠΑ, είναι αρμόδιο να κρίνει τα κράτη-μέλη για θέματα ΚΕΠΑ. Και αν δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αποζημιώσει για, τα, για τις ζημίες που προκάλεσε ε, ένα τάγμα γαλλικό ε, κάπου σε μια χώρα, η Γαλλία είναι υπεύθυνη. Και η απόφαση Ματιού, η σχετική νομολογία, αυτή την ερμηνεία και την απόφαση έδινε. Οπότε θα πρέπει το δικαστήριο να αποφασίσει τι προτιμά. Να ερμηνεύεται και να κρίνεται η ΚΕΠΑ από τα κράτη-μέλη ή να αναλάβει και αυτό τις ευθύνες του για θέματα ΚΕΠΑ. Αυτά ευχαριστώ. Thank uh, ευχαριστούμε πολύ. Ας περάσουμε τώρα στην καθηγήτρια Σόνια Μωράνο Φουαντή, καθηγήτρια νομικής και διευθύντρια στο Κέντρο Νομικής Έρευνας και Πολιτικών Σπουδών, σπουδών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Oxford Brooks, την οποία συνοδεύει ο κύριος Τέλιο Ανδρεδάκη, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ. Από κοινού λοιπόν έχετε κάνει μια παρουσίαση. Κυρία Μωράνο Φουαντή, έχετε το λόγο κυρία Ντανούτα Χούμπνερ, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας να βρισκόμαστε εδώ στην Επιτροπή σας για να μιλήσουμε για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όσον αφορά την μελλοντική πορεία της προσχώρησης αυτής. Θα θέλαμε να επικεντρωθούμε ευθύ αμέσω στα εκκρεμή ζητήματα. Προετοιμάσαμε και μία παρουσίαση PowerPoint, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε την παρουσίασή μας. Δεν ξέρω αν ήδη προβάλλεται. In the meantime, I can continue. Διάμεσο διάστημα θα μπορούσα να συνεχίσω με την παρουσίασή μου. Σήμερα ουσιαστικά θα θέλαμε εμείς να σας παρουσιάσουμε τη δική μας νομική εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με διάφορα εξωτερικά και εσωτερικά σχέδια τα οποία επεξεργαζόμαστε από το 2010 και μετά, τα οποία χρηματοδοτούνται από τη Βρετανική Ακαδημία και από διάφορα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και στόχος ουσιαστικά είναι να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της συνθήκης της Λισαβόνας για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το πιο ενδιαφέρον τμήμα της μελέτης, το οποίο θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε, είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με διάφορες συνεντεύξεις που καταφέραμε να πάρουμε από όλα τα εμπλεκόμενα άτομα στη διαδικασία της προσχώρησης και των σχετικών διαπραγματεύσεων. Ορισμένοι είναι παρόντες σήμερα εδώ και επομένως έχουμε και συνεντεύξεις ή δηλώσεις από τους δικαστές και των δύο πλευρών, και του Δικαστηρίου δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και πριν από μερικές μέρες καταφέραμε επίσης να έχουμε περαιτέρω σχόλια από τους δικαστές των δύο αυτών οργάνων για τα σημαντικά αυτά ζητήματα. Προφανώς εμείς δεν μπορούμε να αρνηθούμε αυτή τη στιγμή ότι δεν περιμέναμε μια τέτοια έκβαση Κατά τη διάρκεια λοιπόν των συνεντεύξεων αυτών, κατά τη διάρκεια τη ίδια τη ακροματική διαδικασία στο δικαστήριο, συνειδητοποιήσαμε ότι το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πάρα πολλέ ανησυχίε, ιδίω όσον αφορά το ζήτημα τη αυτονομία του. Βέβαια γνωρίζουμε ότι οι νομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαπραγματεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο, καθώς επίσης και τα 24 κράτη-μέλη από τα 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν στην όλη διαδικασία, υποστήριξαν το βασικό συμπέρασμα ότι ε, το σχέδιο συμφωνίας προσχώρησης θα έπρεπε να συνάδει με τις ε, συνθήκες. Και η Γενική Εισαγγελέα Κοκότα είπε και η ίδια στις προτάσεις της ότι ε, αν γίνουν οι απαραίτητες τροποποίησεις θα μπορεί αυτό το σχέδιο συμφωνίας να συνάδει με τον ουσιακό δίκαιο. Δεν ξέρω αν μπορούμε τώρα να δούμε τις διαφάνειες της παρουσίασής μας. Πολύ ωραία τις βλέπω. Συνεπώς, Να ξεκινήσουμε από αυτή τη διαφάνεια. Σε ποια σημεία επικεντρωνόμαστε, τι μας απασχολεί όλους ιδιαιτέρως. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να χωρίσουμε την γνωμοδότηση αυτή σε πέντε βασικά θέματα, σε πέντε βασικά ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την αυτονομία, όπως σας είπα. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βρίσκεται πραγματικά στην καρδιά της γνωμοδότησης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτονομία της ένομης τάξης Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτονομία του νοσιακού δικαίου. Το ζήτημα αυτό αναφέρεται συγκεκριμένα σε τρία συγκεκριμένα σημεία της γνωμοδότησης. Το πρώτο έχει να κάνει με τη συμβατότητα σε σχέση με τα δύο αυτά άρθρα τα οποία αναφέραμε, άρθρο 53 της ΕΣΔΑ και άρθρο 53 του χάρτη, το δεύτερο στοιχείο που έχει να κάνει με την αυτονομία και το οποίο εμεί θεωρούμε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω συστάσει είναι το ζήτημα της αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το τρίτο σημείο που έχει να κάνει με την αυτονομία έχει να κάνει με το πρωτόκολλο υπαριθμών 16, ζήτημα το οποίο μπορεί να επιληθεί πιο εύκολα θεωρούμε. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα εκκρεμή ζητήματα τα οποία σε ένα βαθμό συνδέονται με το ζήτημα της αυτονομίας αλλά θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και ξεχωριστά. Άρθρο 344 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και το ζήτημα της αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μηχανισμός παθητικής ομοδικίας, η διαδικασία προηγούμενης εξετάσεως καθώς επίσης και το ζήτημα της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Όπως σας έλεγα λοιπόν, η ε, διατήρηση της αυτονομίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπνοσιακού δικαίου αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο της γνωμοδότησης του Δικαστηρίου. Οι δικαστές ε, στο δικαστήριο έχουν κάνει τις δηλώσεις αυτές που βλέπετε στη διαφάνεια, δηλώσεις που γίνονται στα πλαίσια συνεντεύξεων που πήραμε εμείς θεωρούν ότι πρέπει να είναι οι μόνοι διαιτητές, οι μόνοι ρυθμιστές του ενωσιακού δικαίου και ότι μπορεί να προβλεφθεί μόνο μία πολύ συγκεκριμένη σχέση ανάμεσα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ενωσιακό δίκαιο, ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα κεντρικής σημασίας όσον αφορά τη γνωμοδότηση αυτή. Ουσιαστικά εδώ πέρα δικαστές αναφέρονται στις βασικές αρχές, τα βασικά θεμέλια του ενωσιακού δικαίου. Στη συνέχεια εμείς προσπαθήσαμε να αναλύσουμε το ζήτημα της μη συμβατότητας ανάμεσα στα δύο αυτά άρθρα, άρθρο 53 της ΕΣΔΑ, άρθρο 53 του χάρτη. Είναι πολύ δύσκολο να ζητήσουμε από το δικαστήριο να επαναθεωρήσει την ερμηνεία του άρθρου 53, γιατί η συγκεκριμένη αυτή ερμηνεία προκύπτει από την υπόθεση Μελώνη, και ουσιαστικά συνδέεται με την ίδια την αρχή της αμοιβέ εμπιστοσύνης. Δηλαδή, Πρέπει να δούμε εδώ πέρα σε ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη μπορούν να υπερβούν το ανώτατο επίπεδο παρέμβασης, το ανώτατο επίπεδο προστασίας συγκεκριμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων προβλέπεται από το άρθρο 53 του χάρτη. Αν προβλέπεται ή επιτρέπεται κάτι τέτοιο, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 53 της ΕΣΔΑ, αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια σειρά προβλημάτων, ενδεχομένως να οδηγήσει ακόμα και σε στρεβλώσεις στα πλαίσια του νοσιακού δικαίου. Ακολουθώντας λοιπόν τις δηλώσεις του δικαστηρίου, ξέρουμε βέβαια από τη μία πλευρά ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης και από την άλλη διαπραγματευτές θα είναι κατά τη ίδια τη ιδέα τη τροποποίηση του σχεδίου συμφωνία τη προσχώρηση. Ωστόσο, εμεί πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποιε δυνατότητε να βρεθεί μια πλευρα οτι το συμβουλιο της ευρωπης και απο την αλλη διαπραγματευτε θα ειναι κατα της ίδιας της ιδέας της τροποποιησης του σχεδιου συμφωνιας της προσχωρησης ωστοσο εμεις πιστευουμε οτι υπαρχουν καποιες δυνατοτητες δηλαδή, να δώσουμε μια ξεκάθαρη ερμηνεία των άρθρων αυτών στο σχέδιο συμφωνίας στο δικό μας το έγγραφο, το οποίο απαριθμεί περίπου 15 σελίδες, προτείνουμε και κάποιες άλλες λύσεις, τις οποίες όμως δεν συνιστούμε άμεσα, όπως για παράδειγμα να γίνει μία δήλωση ερμηνείας και να ξεκαθαρίζεται εξ αρχής πώς θα πρέπει να ερμηνεύονται τα δύο αυτά άρθρα. Ενώ μία τρίτη πρόταση ήταν να τροποποιηθεί είτε το ένα από τα δύο άρθρα και τα δύο άρθρα προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν αυτέ τι απαιτούμενε τροποποίησει. Καταλαβαίνετε όμω ότι αυτό είναι μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία που προποθέτει τροποποίηση των ίδιων των συνθηκών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην επόμενη αυτή διαφάνεια αναφερόμαστε στο πρωτόκολλο 16. Το πρωτόκολλο 16 συμφωνήθηκε μετά την σύναψη του σχεδίου συμφωνίας. Επομένως, το πρωτόκολλο 16 δεν αποτέλεσε ζήτημα συζήτησης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Πολλοί στην Ευρώπη είχαν εκφράσει σχετικές ανησυχίες και ουσιαστικά εδώ πρέπει να δούμε ότι το πρωτόκολλο 16 δημιουργεί ένα πρόβλημα σε σχέση με το ζήτημα της άγρας αρμοδίου δικαστηρίου γιατί ενδεχομένως τα ανώτατα δικαστήρια των κρατών μελών να μπορούν να αποφασίσουν να ζητήσουν γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κατά αυτόν τον τρόπο θα παρακάμπτε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 137 όσον αφορά δηλαδή τη διαδικασία του προδικαστικού ερωτήματος, της προδικαστικής παραπομπής και κατά αυτόν τον τρόπο παρακάμπτεται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο. Στο άρθρο 267 ξέρετε ότι υπάρχει συγκεκριμένη υποχρέωση κάθε φορά που προκύπτει ζήτημα ερμηνείας του ενωσιακού δικαίου υπάρχει συγκεκριμένη υποχρέωση παραπομπή στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε όμως ότι αυτό το αποφασίσουν τελικά τα εθνικά δικαστήρια, να πόκειται σε απόφαση των εθνικών δικαστηρίων να χρησιμοποιήσουν το διάβλο αυτό. Θα μπορούσαν ενδεχομένω να ακολουθήσουν κάποια άλλη λύση, κάποιον άλλο δρόμο. Προκύπτει εδώ πέρα λοιπόν ένα ζήτημα περιορισμού της πιθανότητας να χρησιμοποιήσουν τα ανθρώπινα, συγγνώμη, τα νότα δικαστήρια των εθνικών δικαστηρίων το διάβλο αυτό που προποθέτει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρακάμπτοντας κατά αυτόν τον τρόπο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδίως βέβαια όταν προκύπτει ένα ζήτημα με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με την εφαρμογή της ΕΣΔΑ. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει πάλι να έχουμε εδώ πέρα στο σχέδιο συμφωνίας μία ρήτρα, μία διάταξη, στην οποία θα μπορούσε να προβλέπεται απαγόρευση, αν θέλετε, ή να αποθαρρύνονται τα κράτη-μέλη να απευθύνονται και προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ανταυτού να χρησιμοποιούν όντω τη διάταξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νοσιακό δίκαιο όσον αφορά το προδικαστικό ερώτημα από το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσει ο συνάδελφό μου. Όσον αφορά τώρα το άρθρο 33 της Σύμβασης και το άρθρο 344. Για δύο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια που θα είναι ο τελικός ε, ρυθμιστής ε, για να επιληθεί αυτό πρέπει να καταλήξουμε στη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δώσουμε προτεραιότητα στο άρθρο 344 που αφημίζει και λέει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πρέπει να έχει αυτή την ε, νομική αρμοδιότητα. Για να επιληθεί αυτή η τριβή, αυτή η ένταση υπό το πρίσμα μας. Μια εναλλακτική λύση θα ήταν να είχαμε μια δεσμευτική δήλωση υπό το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα ξεκινήσουν οποιασδήποτε προσφυγές κατά του άρθρου 33. Ωστόσο θεωρούμε ότι δεν θα ικανοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με μια τέτοια δήλωση. Η δική μας λύση, η δική μας πρόταση λοιπόν θα ήταν να υιοθετηθεί μια ευρωπαϊκή διάταξη στο σχέδιο προσχώρησης ε, που ρητά θα αποκλείει την αρμοδιότητα υπό το άρθρο 33 του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να επιλύει θέματα τα οποία αφορούν ε, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν πρόκειται για ένα θέμα το οποίο εντάσσεται μέσα στις αρμοδιότητες του ευρωπαϊκού δικαίου. Θεωρούμε ότι αυτή είναι η πιο πρακτικής μορφής λύση που μπορεί να γίνει αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και περνώ τώρα στο επόμενο θέμα, δηλαδή το θέμα των ομοδίκων. Εδώ έχουμε δύο θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Το πρώτο είναι η εμπλοκή της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως ε, συνεναγωμένου και το δεύτερο ο επιμερισμός ευθύνης ε, μεταξύ των του μηχανισμού παθητικής ομοδικίας και των συνεναγωμένων. Εδώ για παράδειγμα όσον αφορά την ίδια την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει κάποια αναθεώρηση από το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αν θα πρέπει ή όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί. Εφόσον επιθυμεί να αποτελέσει μέρος αυτών των εργασιών η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκφράζει την βούλησή της, τότε επαρκεί να έχει το καθεστώς ε, του correspondence, του συνεναγωμένου διότι διαφορετικά αυτό θα παρέβαινε την αυτονομία του ευρωπαϊκού δικαίου και θα θέλαμε να αποφύγουμε μια τέτοια περίπτωση. Όσον αφορά τον επιμερισμό ευθύνη, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αφορά το άρθρο 3 εδάφιο 7 της Συμφωνίας και είναι ένα θέμα που και η γνωμοδότηση και η άποψη του Γενικού Εισαγγελέα συγκλίνουν επ' αυτού. Δηλαδή, είναι προβληματική κατάσταση και προτείνουμε αυτό το τμήμα όσον αφορά την κοινή ευθύνη κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγραφεί, να απαλληφθεί, διότι διαφορετικά θα υπονόμευε την ιδέα του μηχανισμού των, ε, ε, της παθητικής ομοδικίας. Και ένα τελικό θέμα που αφορά τις επιφυλάξεις. Ε, σε, αν σε αυτή τη φάση υπάρχει μια επιφύλαξη που έχει διατυπωθεί σε σχέση με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τότε με βάση αυτή την ε, ε, διάταξη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ειδικό καθεστώς και είναι πάλι μια απόψη επί της οποίας και στη γνωμοδότηση και ο Γενικός σα συνεννούν ότι δηλαδή εδώ έχουμε μια προβληματική κατάσταση που θα πρέπει να αποσαφινιστεί μέσω της επικαιροποιημένης διατύπωσης. Προχωρώντας τώρα στην προηγούμενη εμπλοκή της, Ευρωπα... της προηγούμενης εξέτασης θέλουμε, πρέπει να δούμε κατά πόσο του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Υπό το δικό μας ε, ε, σχέδιο δεν υπήρχε κάποια τριβή. Δέχθηκε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ότι το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όντα ένα εξειδικευμένο δικαστήριο, θα έπρεπε να έχει το τελευταίο λόγο. Αλλά θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει και ερμηνεία εκ προημίου του ευρωπαϊκού δικαίου. Έχουμε λοιπόν κάποιες προτάσεις για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται στην συμφωνία όσον αφορά την ε, προηγούμενη εξέταση, prior involvement, ε, διαδικασία προηγούμενης εξέτασης για την αναζήτηση της της λύσης. Η πρώτη, το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα πρέπει να καταργήσει, να παγώσει τις διαδικασίες σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράσει τη δική της βούληση από πλευράς της να εμπλακεί ως ε, ένας συνεναγόμενος μέσα στο πλαίσιο του μηχανισμού παθητικής ομοδικίας και κάθε φορά που θα υπάρχει μια περίπτωση που θα εμπλέκει το ευρωπαϊκό δίκαιο και θα αποτελεί και θέμα ενδιαφέροντος του δικαστηρίου ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πλήρως να ενημερώνεται ώστε να είναι σε θέση να αποφασίζει αν επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτές τις διαδικασίες και να καταλήξει στον μηχανισμό παθητικής ομοδικίας τελικά. Ε, Πρέπει να υπάρξει λοιπόν αυτή η δυνατότητα ώστε να έχει χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να στοχαστεί και να προβληματιστεί, να δει αν θα επιθυμεί να συμμετάσχει ή όχι σε αυτό το πλαίσιο. Και τέλος το θέμα της αποδοχής του παραδεκτού ε, αυτού του μηχανισμού σε περίπτωση που το δικαστήριο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί. Μόνο το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει αν έχει καλυφθεί ε, και έχει ε, εξεταστεί αυτό το θέμα ή όχι. Και δεν είναι αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να το πράξει αυτό. Και το τελευταίο ζήτημα είναι ότι η ΚΕΠΑ, η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και το θέμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, Mutual Trust, για την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Δυστυχώς δεν ακούγεται το μικρόφωνο της κυρία Παλή. Το θέμα αυτό χαρακτηρίστηκε ουσιώδες. Η έλλειψη δικαιοδοσίας, η περιορισμένη δικαιοδοσία θα προτιμούσα να πω αυτό του δικαστηρίου στο θέμα της κοινή εξωτερικής πολιτικής και κοινή πολιτικής ασφάλειας, της ΚΕΠΑ. Θεωρώ ότι το ζήτημα αυτό είναι μείζον, γιατί το ΔΕ δεν θα επιτρέψει εύκολα στο ΕΔΑ, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να ασχοληθεί με αυτό αυτή την ιδιαιτερότητα. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει το μονοπόλιο σε ό,τι αφορά την εξέταση της νομιμότητας των νομοθετικών πράξεων και έχει περιορισμένη δικαιοδοσία με βάση το άρθρο 215. Οπότε, αν ε, έχουμε ένα νομικό μέτρο που θεσπίζεται από το Συμβούλιο και που περιλαμβάνει κάποια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επηρεάζει φυσικά πρόσωπα, τότε το δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί. Σε άλλες περιπτώσεις όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει αυτή την ε, αρμοδιότητα για την εξουσία. Οπότε κάτι τέτοιο δεν ήταν συμβατό με το θέμα της αυτονομίας και το θέμα του μονοπωλίου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να επιτρέψει στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επιληθεί αυτών των θεμάτων χωρίς το ίδιο το ΔΕ προηγουμένως να μην είχε την ευκαιρία να εξετάσει την υπόθεση. Και αυτό είναι από τα βασικά στοιχεία, ε, τα σημαντικά επιχειρήματα που είδαμε και στο εμπειρικό μας έργο. Εμείς ε, υποβάλλουμε τρεις ε, διαφορετικές προτάσεις, επιλογές που ε, και με την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η πρώτη λύση, απλούστερη ίσως, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλει επιφύλαξη ε, από την ΕΣΔΑ και να εξαιρέσει την ΚΕΠΑ ή να απλουστεύσει το θέμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης για τα θέματα του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Και παρόλο που η Γενική Εισαγγελέα Κόκοτ είπε στην γνωμοδότησή της ότι μία επιφύλαξη που θα αποκλείει την ΚΕΠΑ δεν είναι δυνατή λόγω των κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούνται, αν τελικά τα κράτη-μέλη ή ο διαπραγματευτής τα καταφέρουν να το υποβάλλουν, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την, ομολογία του ΕΔΑ στην περίπτωση Γκράντες και Στίβενς κατά του Ιταλικού κράτους. Οπότε η επιφύλαξη δεν, μπορεί, δεν χρειάζεται να είναι γενικού χαρακτήρα, να είναι γενική επιφύλαξη. Θα μπορούσε να αναφέρει συγκεκριμένα άρθρα των συνθήκων που αφορούν το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και έτσι μπορούμε να είμαστε πιο ειδικοί και πιο συγκεκριμένοι και όχι τόσο γενικοί. Βέβαια υπάρχει και μία αρνητική πλευρά, ένα μειονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι ότι μία επιφύλαξη σε περίπτωση που υπάρχει μια τεράστια επανάσταση του Ευρωπαϊκού Ενωσικού Δικαίου με μελλοντική επέκταση αρμοδιοτήτων, το θέμα της επιφύλαξης είναι σημαντικό. Γι' αυτό προτείνουμε μια δεύτερη λύση την τροποποίηση του σχεδίου συμφωνία προσχώρηση προκειμένου να περιλάβει μια διάταξη που θα αποκλεί το χώρο ελευθερίας, ασφάλεια και δικαιοσύνης και την ΚΕΠΑ από τη δικαιοδοσία του ΕΔΑ, του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και μια διάταξη που θα διευκρινίζει το πεδίο εφαρμογή τη αρχή τη αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και αυτή η λύση βέβαια προσκρούει σε κάποιου περιορισμού, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε δυνητικά μία αναθεώρηση της συνθήκης και τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό το θέμα. Η πρώτη επιλογή που την αισθενίζονται και κάποιοι από τους δικαστές που δεν την κρίνουν ως άμεση λύση αλλά μια μελλοντική θα ήταν και μια αναθεώρηση της συνθήκης προκειμένου να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες και εξουσίες του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Προς το παρόν εμείς προτείνουμε τη δεύτερη λύση που είναι και πιο εφικτή σε αυτή τη φάση. Οπότε, εν κατακλείδη, τα συμπεράσματα θα τα περιγράψει ο συνάδελφος. Εν κατακλείδη, λοιπόν, η γνωμοδότηση 2 του 2013 ήταν πρόσβενη, ευνηδιαστική και κλώνησε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας όλων των ενδιαφερομένων. Μας αναστάτωσε λοιπόν, ιδιαίτερα μάλιστα μετά την θετική γνωμοδότηση της Γενικού Εισαγγελέως, της κυρίας Κοκότ. Η αντίδραση των ακαδημαϊκών ήταν θλίψη και απογοήτευση. Αυτό ακούσαμε από του πανεπιστημιακού. Βέβαια, 16 μήνε μετά, η απογοήτευση έχει μετατραπεί σε προβληματισμό και επικρατεί μεγαλύτερο ρεαλισμό. Αυτό το διαπιστώνουμε. Έχει αλλάξει το κλίμα και φάνηκε και από του προλαλήσαντες. Βρισκόμαστε τώρα σε ένα σταυροδρόμι, σε ένα σημείο καμπής και πρέπει να δούμε την ακολουθητή απορία. Οι πρόεδροι Ισκουρής και Κώστα το 2011 μίλησαν για μια σταδιακή σύγκληση. Δεν θα είναι εύκολη βέβαια η διαδικασία, ούτω ή άλλω. Εξορισμού ήταν δύσκολη η διαδικασία, η διαδικασία τη προσχώρηση. Οπότε η γνωμοδότηση αυτή είναι ένα έλεγχο ε, τη πραγματικότητα. Δεν θα πρέπει να νιώθουμε ούτε συντετριμένοι, ούτε συνταραγμένοι, ούτε αναστατωμένοι, ούτε ε, θλιμμένοι. Η διαδικασία είναι περίπλοκη, φάνηκε αυτό από τη γνωμοδότηση και χρήζει περαιτέρω προσαρμογή. Και για να παρα παραφράσω αυτά που είπε η Γενική Συγγελία Κοκότ, όντω ο διάβολο μπορεί να βρίσκεται στι λεπτομέρειε. Και αυτό το διαπιστώσαμε και με την κατάσταση αυτή. Οπότε να και στα ενδιαφερόμενα μέρη να κρίνουν ποια είναι η πιο κατάλληλη ακολουθητέα πορεία. Γιατί χρειάζεται στι ε, μελλοντικέ διαπραγματεύσει ε, μια άλλη προσέγγιση και μεγαλύτερο ρεαλισμό. Γιατί ε, δεν αρκούν μόνο οι νομικέ λύσεις, χρειάζεται και πολιτική βούληση από τα κράτη-μέλη, από τις κυβερνήσει για να εφαρμόσουν τη συμφωνία και να, την, και να λειτουργήσει και στην πράξη. Είμαστε αισιόδοξοι πάντω. πιστεύουμε ότι είναι δυνατό κάτι τέτοιο, άλλωστε το προβλέπουν και οι συνθήκες, είναι υποχρεωτικό και ακόμη και αν είναι χρονοβόρη διαδικασία πιστεύω ότι τελικά θα αποβεί προ όφελο των Ευρωπαίων πολιτών ε, γιατί ενισχύεται το επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό είναι το ζητούμενο που θα πρέπει να αποτελεί και το φάρο των προσπαθειών μας. Και σας ευχαριστούμε θερμά που μας υποδεχθήκατε στην ακρόαση. Ευχαριστούμε και εμείς. Περνάμε τώρα στη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε τον Διευθυντή Ρικάρντο Πάσους που είναι Διευθυντής Θεσμικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ, Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν γνωρίζω αν έχουμε πάει πολύ πιο πέρα από αυτά τα οποία συζητήσαμε την τελευταία φορά κατά τον Φεβρουάριο εφέτος, 26 Φεβρουαρίου. Πολλά συντάχθηκαν από πλευράς μας όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Όμως ένα ή δύο θέματα ο καθηγητής Ζακέ θα μπορέσει ίσως να διαφωνήσει που βρίσκονται υπέρ αυτής της νομικής ε, γνωμοδότησης. Όλες οι άλλες τοποθετήσεις ήταν ε, ε, κατά και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το ιστορικό η προσχώρηση δεν είναι μόνο αποκλειστικά νομικού χαρακτήρα. Φυσικά πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 εδάφιο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που εκφράζονται υπό το πρωτόκολλο 8. Όμως η όλη διαδικασία του να υπάρχει ένας διεθνής έλεγχος και η συνολική ιδέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο ε, που δεν θα έχει την ε, τον τελευταίο λόγο για τα δικαιώματα του ανθρώπου έχει πολιτικές επιπτώσεις. Αυτό το κατανοούσαμε ευθύ εξ αρχής αλλά και τα ίδια τα κράτη-μέλη όταν δέχθηκαν την αρμοδιότητα, την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το έπραξαν αυτό Κατά τη διάρκεια ερωτημάτων που ανεφύησαν, παράδειγμα, γιατί να μην αναμείνουμε μέχρι ότου να διευθετηθούν τα πάντα, άπαντα τα θέματα και μετά να διαπραγματευτούμε το θέμα της προσχώρησης. Θέματα, για παράδειγμα, της ε, αρμοδιότητας ε, του πρωτοδικείου ή της του, πρώτου επίπεδου. Ε, αυτό ακριβώς ήταν εκείνο το οποίο για πολλές ε, χώρες ε, που οδηγήθηκαν στο να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προς όφελος της Δημοκρατίας η Πορτογαλία για παράδειγμα όταν προσχώρησε σε αυτή τη σύμβαση η Πορτογαλία το 1976 προσχώρησε σε αυτή τη σύμβαση Φυσικά είχε συνδυτοποιήσει η πορτογαλική κυβέρνηση ότι θα υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με νομικά θέματα όσον αφορά το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τα πορτογαλικά δικαστήρια. Η Γαλλία, η Γαλλία δέχθηκε μόνο την ε, αναγνώριση της ε, νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από πλευράς ε, του Υπουργού Δικαιοσύνης ε, και του Πρωθυπουργού έγινε αυτό το διάβημα αλλά πήρε χρόνια πολλά, ολόκληρα χρόνια για την ε, Γαλλία για να οριμάσει αυτό το θέμα. Έχει λοιπόν και ένα πολιτικό, μια πολιτική συνιστό σε αυτό το θέμα. Αυτό όμως πολλές φορές ε, το αμελούμε σε αυτή τη συζήτηση παρότι έχει τη σπουδαιότητά του. Ας αναφερθώ σε ένα άρθρο, εξαιρετικό άρθρο ε, ενός καθηγητή που αναφέρεται στο ζήτημα αυτό και που λέει ότι ο λόγος, ο στόχος της προσχώρησης είναι να μπορέσουν ε, να ε, συνάδουν τα θέματα αυτά όσον αφορά τα θέματα παραβίασης ε, δικαιωμάτων από, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήταν συγχωρητέο να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα αυτή η άποψη έχοντας γνώση της τοποθέτησης γνωμοδότησης όσον αφορά την αναφορά αυτού του στόχου για την ενίσχυση της θεμελιώδους προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου για τους πολίτες. Και αληθεύει, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτή την προοπτική, ότι κάνουμε λόγο για ανθρώπους εδώ, για πολίτες και την προστασία των ατομικών αυτών δικαιωμάτων των πολιτών αυτών και όχι τόσο ε, θέματα για θέματα μεταξύ αρμοδιοτήτων, μεταξύ δικαστηρίων. Και αυτό είναι ακριβώς ε, το θέμα στο οποίο πρέπει να εστιαστούμε σε αυτό το ζήτημα. Για το ποιο θα έχει τον τελευταίο λόγο, για παράδειγμα, σε σχέση με την παραβίαση δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα είναι το, το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο, ε, είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο ε, Λουξεμβούργο, θα είναι το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Ποιο θα έχει τον τελευταίο τελευταίο λόγο για όλα αυτά. Υπήρξε και κάποια έκπληξη για την γνωμοδότηση επειδή το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το γνωρίζει αυτό η Επίτροπη και ε, η ίδια είχε εμπλακεί κατά τη διάρκεια των διαδικασιών και διαβουλεύσεων και είχαν ε, προταθεί και κάποια θέματα μένοντας και επιμένοντας στο μηχανισμό προηγούμενης συμμετοχής εδώ όμω, σε σχέση με τον μηχανισμό prior involvement mechanism υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση ε, αφορώνται και που ε, δεν ε, πρέπει να διαφύγουν της προσοχής των διαπραγματευτών και σε σχέση με το πόσο έχουμε προοδεύσει δεν μου φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος σε σχέση με την προηγούμενη τάξη πραγμάτων όπως τα είχαμε συζητήσει κατά το παρελθόν. Σε κάποια υστερότερη φάση θα πρέπει να υποβάλει ε, κάποιες κατευθυντήρες γραμμές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε στην επαναδιαπραγμάτευση αυτού του θέματος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο σε κάποια άτυπη βάση. Σε κάποια υστερότερη φάση θα πρέπει πρέπει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώσει τις ε, διαπραγματευτικές εκείνες συστάσεις και οδηγίες που έχει να προτείνει προς το Συμβούλιο για τη διαπραγμάτευση και να τις ε, αναπέμψει και προς το Κοινοβούλιο προς εξέταση. Ε, σε αυτή τη φάση ίσως θα μπορέσουμε να δούμε πιο συγκεκριμένα, πιο χειροπιαστά, με μεγαλύτερη σαφήνεια πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προχωρήσει. Και νομίζω χρειαζόμαστε να, έχουμε αυτό το κείμενο τότε ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν με τον πιο σωστό τρόπο. Ένα πράγμα όμως είναι βέβαιο και πιστεύω ότι και εδώ θα πρέπει να αποτίσω φόρο τιμή παρεμβάσεις που έγιναν από πλευράς των καθηγητών και του καθηγητού Ζακέ σήμερα το πρωί είναι τουλάχιστον σαφές ότι υπάρχουν δύο μίζωνα ζητήματα τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Το θέμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και το ζήτημα της ΚΕΠΑ. Για την αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς την υφή του προβλήματος. Ωστόσο όμως για την ΚΕΠΑ τα πράγματα είναι ακόμα δυσχερέστερα ίσως. Θα μπορούσα να συμφωνήσω με την καθηγήτρια Σόνια Μοράνο για την ιδέα που προτείνει κάποια ένσταση ή επιφύλαξη για την ΚΕΠΑ. Νομίζω ότι νομικά και πολιτικά κάτι τέτοιο θα ήταν απαράδεκτο. Το Κοινοβούλιο επέμεινε στην ε, ιδέα του να υπάρχει η νομολογία του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τα θέματα της ΚΕΠΑ γνωρίζοντας όμως ότι το ε, δικαστήριο του Λουξεμβούργου δεν είχε αρμοδιότητες για θέματα ΚΕΠΑ. Εδώ όμως αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει μια πρόσθετη αξία για την ε, νομική προστασία άτομα δηλαδή ή σε σχέση με την Ένωση για τα θέματα της ΚΕΠΑ θα μπορούσαν να, να ε, οδηγήσουν σε αυτή την κατεύθυνση εμπλουτίζοντας τις, τα πλαίσια. Όμως το δικαστήριο ανέφερε ότι από πλευράς αναθεώρησης, από πλευράς ΕΕ και ε, ε, ε, υπό το πρίσμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν μπορούν να αναφέρονται αποκλειστικά σε ένα δικαστήριο, διεθνές δικαστήριο το οποίο θα βρίσκεται εκτός νομικής δομής και αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αποκλειστικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού δικαίου όσον αφορά ε, τα θέματα που αφορούν την ε, ΚΕΠΑ μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το επιχείρημα, τα επιχειρήματα αυτά και οι ενστάσεις αυτές είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Είναι όμως επίσης δύσκολο να γίνουν απόλυτα κατανοητά όλα αυτά, διότι όταν έχουμε τα κράτη-μέλη που σε σχέση με το άρθρο 6.2 της νέας συνθήκης όταν συντάχθηκε αυτό γνώριζαν τα κράτη-μέλη ότι η προσχώρηση ήταν υποχρεωτική σε σχέση με το άρθρο 6.2 και γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν ήταν αρμόδιο για τα θέματα της ΚΕΠΑ. Δεν νομίζω ότι το έπραξαν αυτό επειδή δεν είχαν συνειδητοποιήσει το τι συνέβαινε ήταν αυτονόητο ότι θα, το, το δικαστήριο ε, θα μπορούσε να έχει την αρμοδιότητα ότι παρότι το δικαστήριο δικαιωμάτων ανθρώπου μπορεί να μην ήταν αρμόδιο για τα θέματα αυτά και το κοινοβούλιο όπως αναφέρθηκε στο ψήφισμά του στη, στο ψήφισμα 17η Μαΐου 2010 ότι η προσχώρηση θα αντισταθμίζει το γεγονός ότι θα είναι πιο περιορισμένο το φάσμα μα αυτό παρέμβασης εμπλοκής όσον αφορά την ΚΕΠΑ προσφέροντας την δικαστική εκείνη εποπτεία που θα απαιτείται. Από πλευράς του Γενικού Εισαγγελέα καταδείχθηκε ε, μεγάλη κατανόηση για αυτό το θέμα και αναφέρθηκε ότι η νομική προστασία των πολιτών δυναμώνεται και δεν αποδυναμώνεται δεδομένης μιας τέτοιας κατάστασης αν, καθώς αναγνωρίζεται η διεθνής δικαιοδοσία. Θα πρέπει να αναμείνουμε λοιπόν να υπάρξει η δημιουργική πρωτοβουλία με φάνταστο τρόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διευθετηθεί αυτό το θέμα με την προσπάθεια πρότασης μιας λύσης που θα μπορούσε να είναι αποδεκτή. Δεν απορρίπτω απόλυτα την ιδέα μιας ε, επιφύλαξης ή ένστασης αν όμως θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια αναθεώρηση της ηθίκης, αυτό θα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και θα πρέπει να είναι σαφές για το δικαστήριο του ανθρώπου, το, το, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι αν διασφαλίζεται αυτή η αρμοδιότητα τότε το θέμα θα, θα έχει διευθετηθεί. Πρέπει να δούμε τα θέματα λοιπόν ΚΕΠΑ και συμφωνώ υπό αυτό το πρίσμα με τον καθηγητή Ζακέ, αυτό απαιτεί και κάποιο χρόνο που πρέπει να αναλωθεί για να καταλήξουμε σε μια διευθέτηση. Προσβλέπω στο, να δω και αδειμονώ να δω πώς θα προβεί στην ε, πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται αυτή τη στιγμή να ικανοποιήσει αιτήματα από όλε τι πλευρέ. Δεν ξέρω πώ θα τα καταφέρει. Ας α, περάσουμε στον τελευταίο μιλητή. Λογικά προβλεπόταν ο κύριος Κλοντ Μωράες, επικεφαλής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων. Δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει, διότι έχουν πάρα πολλά ζητήματα προς εξέταση στη δική του Επιτροπή. Επομένω, η κυρία Μπάρμπαρα Σπινέλη, αντιπρόεδρός μας, θα παρουσιάσει την άποψη του κυρίου Κλοντ Μωράες, εξ ονόματος Επιτροπής του. Ένας από τους πρόεδρους μου, σε ευχαριστώ Ντανούτα, μου ζήτησε να παρουσιάσω τη δική του την άποψη. Αναφέρομαι βέβαια στον Κλοντ Μωράες, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, αγαπημένοι προσκεκλημένοι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για την ε, δυνατότητα που μου δίνει να συμμετέχω στην πολύ σημαντική αυτή δημόσια ακρόαση και Ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος του κύριου Κλωτ Μωράης, ο οποίος δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. Αυτή τη στιγμή προεδρεύει μια συνεδρίαση σε Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και όπως είπε και η Πρόεδρός μας θέλει από μένα παρουσιάσω την δική του την άποψη. Η προσχώρηση Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί προφανώς υποχρέωση προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωση και απαιτείται προκειμένου να έχει το δικαστήριο ένα επιπλέον μηχανισμό για την καλύτερη προστασία και εφαρμογή της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά αυτόν τον τρόπο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα λογοδοτούν ακόμα περισσότερο για τις πράξεις τους ή τις παραλήψεις τους σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Συνεπώς, θα πρέπει η προσχώρηση αυτή να λάβει χώρα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο, μάλλον ακριβώς αυτό είπανε τα κράτη-μέλη στο ψήφισμα του Σεπτεμβρίου του 2015 όσον αφορά την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είπε και το Κοινοβούλιο μέσω της έκθεσης Φεράρα. Είναι πολύ σημαντικό το, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ιδίω στον τομέα των πολιτικών ελευθεριών, όσον αφορά δηλαδή την κράτηση, το ποινικό δίκαιο, όσον αφορά την προστασία ιστοτικής ζωής, όσον αφορά την ε, μεταφορά, μυστική μεταφορά κρατωμένων από τη CIA και ιδίω όσον αφορά την ομολογία στον ε, τομέα του ποινικού δικαίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η αρχή της αμοιβέ εμπιστοσύνη και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω μιας υψηλότερης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς αυτό, η νομολογία του ε, Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπνέεται από την ομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου με έναν τρόπο ιδιαίτερα επικοδομητικό, μέσω δηλαδή ενός επικοδομητικού διαλόγου, ο οποίος ίσχυε στο παρελθόν και πρέπει να συνεχιστεί. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ανέκαθεν ζητούσε την, εσχύση, την ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωτών δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη μέσω συγκεκριμένων εργαλείων. Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω της χρησιμοποίησης και του μηχανισμού παθητικής ομοδικίας αποτελεί ένα τέτοιο εργαλείο. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, μεταξύ άλλων, ζητά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση να πράξει σωστά τη δουλειά της και τα καθήκοντά της και να δημιουργήσει ένα νέο μηχανισμό μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται η συμμόρφωση όλων των κρατών μελών με τις κοινέ αρχές που έχουμε στο άρθρο 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά αυτόν τον τρόπο θα θεραπεύονται τα εφιστάμενα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει. Η Επιτροπή μας αυτή τη στιγμή προσπαθεί να συντάξει μαζί με την Επιτροπή ΑΦΚΟ μία σχετική εισήγηση, έκθεση, με τη συνεργασία του κυρίου Σόπφλιν, μέσω της οποίας θέλουμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια νέα νομοθεσία για τη δημιουργία ενός μηχανισμού για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη θεμελιώδη δικαιώματα. Και μέσω του μηχανισμού αυτού όλα τα κράτη-μέλη θα συνάδουν με την συνθήκη και με το χάρτη, ιδίω όσον αφορά την προστασία των θεμελιών δικαιωμάτων μέσω κοινών αρχών και κοινών δικτών. Επί του παρόντος, αν ένα κράτος μέλος φαίνεται να παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορεί τελικά να υποχρεωθεί, μάλλον, μπορεί τελικά να βρεθεί σε μια κατάσταση όπου είτε παραβιάζει το νοσιακό δίκαιο προκειμένου να σεβαστεί την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, το αντίστροφο, να παραβιάσει τελικά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκειμένου να συνταχθεί, να συμμορφωθεί με το νοσιακό δίκαιο. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να βρεθούν συγκεκριμένε λύσει όπω στην υπόθεση Μάριου που είχε να κάνει με το δικαίωμα να ψηφίζουν για τι ευρωπαϊκέ εκλογέ και οι πολίτε που διαμένουν στο Γεβραλτάρα. Διαφοροποιείται η κατάσταση όταν ε, τα όσα προβλέπονται στο χάρτη συνάδουν με τα όσα προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όταν έχουμε δηλαδή η ίδια παρενθερή άρθρα με διαφορετική όμως ερμηνεία. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στο χάρτη για συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά για παράδειγμα το ζήτημα του ασύλου ή το ζήτημα των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. Έχουμε δηλαδή στο χάρτη κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να μην προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο χάρτης λοιπόν είναι αυτόνομος, περιέχει πολλές φορές διατάξεις που υπερβαίνουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά έχει και ένα περιορισμένο πεδίο εφαρμογή. Αυτό μην το ξεχνάμε. Εν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι μολονότι υπήρξαν διάφορες αντιδράσεις σε σχέση με την γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιδράσεις οι οποίε ήταν αρκετά απεσιόδοξε, Υπό το φω όμως και τη σημερινή ε, ανταλλαγή απόψεων, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρεί ότι πρέπει να σημειώσουμε αυτή τη στιγμή πρόοδο, πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο, προκειμένου να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία στη διάθεσή μα για να εφαρμόζονται για όλου του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα ανθρώπινα δικαιώματα όπω αυτά προβλέπονται από τι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Θα ακολουθήσει η συζήτηση. Μην ξεχνάτε ότι δεν είμαστε εδώ για διαπραγματεύσει, αλλά για ανταλλαγή απόψεων. Και όλε οι προτάσει είναι πρόσδεκτε και τα σχόλια που τροφοδοτούν και εμπλουτίζουν τη συζήτηση επίση ευπρόσδεκτα. Και δεν εννοώ μόνο τα σχόλια των εκπρόσωπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Ραμόν Χαουρέγγι είναι ο πρώτο ομιλητή που ήταν ο εισηγητή τη ΑΦΚΟ για την έναρξη τη διαδικασία προσχώρηση Ευρωπαϊκή Ένωση στην ΕΣΔΑ. Ραμόν, σε ακούμε. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ισπανικά, φορέστε τα ακουστικά σα αν θέλετε να με καταλάβετε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τις ομιλίες σας, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, ε, περίπλοκες, διαφωτιστικές και μου δημιούργησαν ε, μια διπλή ανησυχία. Καταρχήν, διαπιστώνω ότι η διαπραγματεύση Πραγματεύσει από το Φεβρουάριο του 2015. Ο Ρικάρτο Πάσο μιλούσε για το Φεβρουάριο, αλλά ποιο Φεβρουάριο, ποιο χρόνο. Φέτος, πέρυσι. Γιατί την πρώτη ακρόση την είχαμε το Φεβρουάριο του 2015, αν δεν κάνω λάθος. Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος δηλαδή που είχαμε συνεδρίαση για το ίδιο θέμα και είχαμε αναλύσει την απόφαση του Δεκεμβρίου του 2014. Και Δεν βλέπω ιδιαίτερες εξελίξεις στο τελευταίο χρόνο. Εγώ πρόοδο δεν είδα, απλώ διαπιστώνουμε ε, την ίδια κατάσταση και συγκρίνω τις σημειώσεις μου από την ακρόαση του προηγούμενου χρόνου και βλέπω ότι ε, και σήμερα ακούσαμε τα ίδια επτά προβλήματα. Τα πιο σοβαρά είναι η ΚΕΠΑ και η αμοιβέμπιστοσύνη εμπιστοσύνη και τα άλλα πέντε λιγότερο σοβαρά. Αλλά αυτά τα σημεία είναι τα προσκόμματα και είναι τα ίδια από πέρσι. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή τίποτα. Επίσης, ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης διαπίστωσε ότι τα κράτη-μέλη του περιμένουν τις νέες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συζητηθούν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Οπότε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι από το Δεκέμβριο του 2014, που είχαμε την περίφημη απόφαση, την περίφημη γρομοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μέχρι σήμερα, απλώς περιοριζόμαστε στη διαπίστωση της τεράστιας δυσκολίας ανέβρεσης ε, διεξόδου στο πρόβλημα. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου αντίληψη. Και φυσικά σας μιλάω για μια περισσότερο πολιτική παράνομική λύση γιατί είμαστε μάρτυρες μιας συζήτησης μεταξύ νομομαθών, αλλά εμείς είμαστε εκπρόσωποι, πολιτικοί, ακόμη και αν έχουμε σπουδάσει νομική, δεν έχουμε την ικανότητα και την ε, ε, κριτική ανάλυση που μπορείτε να κάνετε εσείς. Και αυτό με οδηγεί στα εσείς εξής δύο σκέψεις που πρέπει να δούμε ως ζητήματα. Το πρώτο, λαμβάνοντας υπόψη ότι πιθανότατα το πολιτικό κλίμα στο οποίο ζούμε μας παρουσιάζει δύο σημεία αναφοράς που ακόμα πιο σημαντικό καθιστούν για τους Ευρωπαίους πολίτες στην προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη σύμβαση. Πρώτον, επειδή ήδη διαπιστώνεται στην πολιτική συζήτηση του σώματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η αμφιβολία ή αμφιβολίες που δημιουργούνται για την υλοποίηση και την εφαρμογή, την συμμόρφωση με τα δικαιώματα του ανθρώπου από πλευράς κρατών μελών. Και όλο και πιο συχνό είναι το ζήτημα το οποίο αφορά την, τον επιμερισμό των, ε, των εξουσιών στα κράτη-μέλη, στα κράτη-μέλη σε σχέση με το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών που φυσικά εξακολουθεί να υφίσταται ο χώρος προστασίας που τα κράτη-μέλη τα οποία ανήκουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης δημιουργούν και έχουν λόγω του ότι είναι κράτη-μέλη. Υπάρχει όμως και η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το αν σε σχέση με τα, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς επίσης και η συζήτηση για την ελευθερία που διεξάγεται στη συζήτηση. Ζούμε μια πολύ ευαίσθητη στιγμή στην Ευρώπη και τα επόμενα 20 χρόνια στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα έχουμε τεράστιες τριβές ε, όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και όλα αυτά. Και πράγμα που καταδεικνύει σφαιρικά και συνολικά ότι η προσχώρηση ότι όταν συμφωνήσαμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνα θα συμπεριλάμβανε την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωση, αυτή η αρχή τη της διπλής προστασίας των Ευρωπαίων πολιτών έχει κάθε φορά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Αυτή είναι η διαπίστωση στο πολιτικό πλαίσιο. Και σε αυτό το πλαίσιο έχω μία ερώτηση και μία πρόταση. Η ερώτηση που αφορά τους εκπροσώπους τη Προεδρίας της Προεδρίας της Ένωσης, αυτή τη στιγμή δηλαδή του Συμβουλίου, ποια είναι η άποψη των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα ζούμε σε αυτή τη συγκυρία δύσκολες στιγμές όσον αφορά την διαπραγμάτευση του θέματος της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου την Ευρωπαϊκή Ένωση του Brexit και έχουμε διαπραγματεύσει σε ποια είναι η άποψη των κρατών μελών, ποιες είναι οι απόψεις των κρατών μελών σε σχέση με τα θέματα που τίθεται υποσυζήτηση. Διότι ένα θέμα είναι να εκπονεί τεχνικές προτάσεις η Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Επιτροπή σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπή και άλλο θέμα είναι το τι συμβαίνει με τα τα κράτη-μέλη και το πώς θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ερώτημα, ποια είναι εδώ η λειτουργία τους και η τοποθέτησή τους, διότι είδα από μία από τις παρατηρήσεις ε, του Νομοσυμβούλου του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι είπε προσοχή, μην κάνετε τροποποιήσεις στη, συμφωνία στο ένα ή άλλο σημείο, διότι δεν θα το δεθούν αυτό τα κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πράγμα που με κάνει να, να αντιλαμβάνομαι ότι από πλευρά του Συμβουλίου της Ευρώπης υπάρχει μια πολύ αμυντική τοποθέτηση όσον αφορά μια πιθανή τροποποίηση της συμφωνίας που δεν θα την ε, αποδεχόντουσαν καθόλου εύκολα. Και για να ολοκληρώσω Πρόεδρε, διερωτώ με αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει να πει κάτι και μπορούσε να πει κάτι. Είχαμε αναφέρει το ότι δεν είναι απλά και μόνο έκφραση βούλησης ή προσχώρηση. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά νομικών ε, διατυπώσεων ε, υπέρ και η ερώτηση τώρα που τίθεται είναι δεν θα έπρεπε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να μπορέσουμε να διατυπώσουμε κάποια πράγματα σε σχέση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο εκφράζοντας τη βούλησή μας από πλευράς μας ότι θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και ότι πρέπει να διευθετηθεί. Αυτή θα ήταν η πρότασή μου σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε, Ραμόν. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Ντανούτα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μας, γιατί πραγματικά οι παρουσιάσεις τους ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Υπάρχει ένα ζήτημα όμως, επί του οποίου θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα και πιο συγκεκριμένα έχει να κάνει με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και η σχετική απόφαση που έχει λάβει το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν είναι αν η απόφαση αυτή του Δικαστηρίου αποτελεί κατά κάποιον τρόπο ένα μήνυμα, πώς να το θέσω, ένα έμεσο μήνυμα, ένα κωδικοποιημένο μήνυμα, το οποίο μας αποστέλει το δικαστήριο προς εμάς, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και προς τα υπόλοιπα δικαστήρια. Επί της ουσίας, τι θέλω να πω. Αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι αν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επιλύσουν το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει, έλλειψη δηλαδή αρμοδιότητας όσον αφορά το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ζητήματα κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Υπάρχει μια έλλειψη αρμοδιότητα του δικαστηρίου ω προ αυτό. Στην πράξη, ελλείψη τέτοια αρμοδιότητα καλούμαστε εμεί οι πολιτικοί να αναλάβουμε δράση, θεωρώ. Θεωρώ ότι εμεί θα πρέπει να δώσουμε αυτή την αρμοδιότητα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένω, αυτό είναι το μήνυμα το οποίο προκύπτει από την απόφαση του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν υπάρχει τελικά μια τέτοια έκκληση, αν υφίσταται μια τέτοια έκκληση προ εμά του πολιτικούς και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμεί τι κάνουμε. και ο κύριος Πάσος και άλλοι ομιλητές έχουν απόλυτο δίκιο όταν λένε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει επιτέλους να αναλάβει δράση μετά από όλες αυτές τις διατοχικές δημόσιες ακροάσεις που είχαμε για αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει ειλικρινά να τροποποιήσουμε τελικά τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διερωτάμε ειλικρινά, για ποιο λόγο να τροποποιήσουμε τις συνθήκες, εφόσον ήδη υφίσταται ένα άρθρο της συνθήκης στο οποίο προβλέπεται η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προφανώς προκύπτουν επιμέρους νομικά προβλήματα, αλλά διερωτάμε, δεν ξέρω αν θα μπορούσατε εσείς να μου πείτε πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τις διαπραγματεύσεις προτού να προκύψει μία τροποποίηση της συνθήκης αν αυτή κρυθεί τελικά αναγκαία. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό θα ήθελα να θέσω και άλλα ερωτήματα, αλλά νομίζω ότι ήδη μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Μην ανησυχείτε, μπορείτε και στη συνέχεια να προσθέσετε κάποιο σχόλιο. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος από τους συναντέρφους να λάβει το λόγο. Γιατί αν θέλει κάποιος άλλος από την ομίγυρη να υποβάλει ερωτήσει, να κάνει σχόλια, Άντριου, εγώ σε προκάλεσα. Ο κύριος Άντριου Νταφ. Θα ήθελα να πω σε σχέση με την εκστρατεία που γίνεται για το Βρετανικό δημοψήφισμα. Το ζήτημα του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, αναδείχθηκε ως ε, αρκετά επίμαχο. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ θα πρέπει να υιοθετήσει όσο πιο επικοδομητικό ρόλο γίνεται και όσο πιο θετικό ρόλο γίνεται και να προσπίσει και να προωθήσει το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Αυτός ο θετικός και επικοδομητικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερος ε, σημαντικός. θα πρέπει να υστερεί σε σχέση με τις προσδοκίες ε, που είχαμε κατά την εκπόνηση, κατά την κατάρτιση του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και δόθηκε, ε, ελυθή απόφαση να δοθεί ε, με τη δεσμευτική ισχύ του, δεσμευτική του χάρτη στο ε, στη συνθήκη της Λισαβόνας και το αντάλλαγμα ήταν η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη ε, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και αυτό δεν πρόκειται να λυθεί μόνο από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο ή το, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο, ή να αντιμετωπιστεί ως ε, ίσονο σημασίας δευτερεύων ή παρεμπίπτων ζήτημα. Το θέμα της αμοιβέ εμπιστοσύνης δίνεται και οφείλει να διευθετηθεί από μια άλλο και μεγαλύτερη σύγκληση μεταξύ των δύο δικαστηρίων. Το θέμα της ΚΕΠΑ μπορεί να διευθετηθεί ικανοποιητικά μόνο με αλλαγή του πρωτογενούς δικαίου προκειμένου να επεκταθεί η δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να καλύπτει όλες τις πτυχές της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμπεριλάβει και αυτό το σημείο στο κατάλογο των ετοιμάτων που καταρτίζει. για τις ε, μελλοντικές αλλαγές στη συνθήκη. Ευχαριστώ, Άντριου. Ε, έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι θα το βάλουμε στην έκθεση Verhofstadt και ελπίζω να είναι θετική η έκβαση και στην ΑΦΚΟ σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία επί της εκθέσεως αυτής. Και επανέρχομαι στους καλεσμένους μας. Ποιος θέλει το λόγο παρακαλώ ο Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας, ο κ. Πάσος. Ευχαριστώ. Να σχολιάσω τις τελευταίες παρατηρήσεις του κυρίου Άντριου Νταφ, που με ιδιαίτερη χαρά τον ξαναβλέπω, για τις αλλαγές στη συνθήκη, ώστε να διευρυνθεί η δικαιοδοσία του ΔΕ για την ΚΕΠΑ. Αν γίνει η αναθεώρηση της συνθήκης, το δικαστήριο δεν έχει λόγο να το θεωρεί ως πρόσκομα αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα περιορίσει τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δείξει μια δημιουργικότητα, μια ευρηματικότητα και να προτείνει άλλη λύση. Ο καθηγητής Ζακέ εργάστηκε στο Συμβούλιο για πολλά χρόνια και είπε ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα να δώσουν δικαιοδοσία ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για θέματα κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Οπότε, αν το Κοινοβούλιο από τώρα σε ένα ψήφισμα ε, ζητήσει ρητά αναθεώρηση της συνθήκης προκειμένου να επεκταθεί η δικαιοδοσία του ΔΕ και σε θέματα ΚΕΠΑ, ίσως ε, έμεσα αποκλείσει άλλους τρόπους για να υπερβούμε το πρόβλημα, να το υπερκεράσουμε. Αυτό θα ήθελα να σας επισημάνω. Ευχαριστώ. Thank you very much, Madam Chair. Ο κύριος Δεγκράβ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χάουρεγγι για την ερώτηση που υπέβαλε προς το Συμβούλιο. Ρώτησε τι κλίμα επικρατεί στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω με τρεις απαντήσεις. Καταρχήν, ισχύει η νομική υποχρέωση προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το θέμα αυτό συζητήθηκε στις 9 Οκτωβρίου πρόσφατα από τους ε, Υπουργούς Δικαιοσύνης και οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν ε, τη δέσμευσή τους ε, υπέρ της, προσ... της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προβλέπουν οι συνθήκες. Και δεν συμφωνώ ότι τίποτα δεν έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο. Έχουν γίνει πολλές τεχνικές συζητήσεις για τα πιο τεχνικά, δικονομικά ζητήματα με βάση τις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα συνεχίσουμε τις τεχνικές συζητήσεις στην αρμόδια ομάδα εργασίας την επόμενη εβδομάδα. Και όπως είπα και προηγουμένως, το Συμβούλιο έχει διατρανώσει τη δέσμευσή του να επιλύσει τις εκκρεμότητες, κυρίως το, ως προς την ΚΕΠΑ και την αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατά προτεραιότητα μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κάτι καινούριο για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Ντεγκράβ. Ο κύριος Πολακέβιτς. Εγώ έχω μια ερώτηση προς όσον αφορά τη στάση του Συμβουλίου της Ευρώπης και των κρατών μελών. Φυσικά λένε ότι δεν μπορούν να ομιλήσουν εξ ονόματος των μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης επειδή δεν έληφθη κάποια πολιτική απόφαση που να έχει ληφθεί από τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης εκτός από την επανάληψη της δέσμευσής τους να, μπορέσει να, να μπορέσουν να ολοκληρώσουν αυτή τις, ε, αυτές τις ε, μέσα στο πλαίσιο το οποίο έχει καθοριστεί. Ωστόσο όμως έχω αποκομίσει την εντύπωση ότι σε σχέση με την ε, συμφωνία προσχώρησης δεν είναι επιθυμητές κάποιες αλλαγές και σε σχέση με τις γραπτές παρατηρήσεις, έντυπες παρατηρήσεις. Η ανησυχία μου σε σχέση με αυτό είναι ότι εντάξει μπορεί κάτι ίσως ε, να τροποποιηθεί, βρισκόμαστε στη διαπραγμάτευση ακόμα. Ωστόσο από πλευρά του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν υπάρχει κάποια νέα εντολή και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις σε αυτή τη χρονική στιγμή και η Συμφωνία Προσχώρησης αποτελεί και αυτή αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Και το μήνυμα τώρα το οποίο θα μπορέσει να αποσταλεί ιδιαίτερα σε σχέση με εκείνα τα σημεία τα οποία καλύτερα θα μπορούσαν να ρυθμιστούν με κάποιους κανόνες ή κανονισμούς ή με κάποια γραπτή δήλωση, ιδιαίτερα όσον αφορά τον εσωτερικό συσχετισμό και σε σχέση με τα θέματα τα ευρωπαϊκά, υπάρχει ίσως και κάποια, ας το πω αμφισβήτηση ή κάποια δυσπιστία σε σχέση με τα κράτη-μέλη όσον αφορά το δικαστήριο δηλαδή υπό το πρίσμα της ε, ε, συνθήκης όταν ε, ε, τίθεται το θέμα της συμφωνίας προσχώρησης πρέπει να δούμε σε σχέση με μια διεθνή συμφωνία το πλαίσιο το οποίο τίθεται σε σχέση με το δικαστήριο του Στρασβουργού και το δικαστήριο του Λούξεμβουργού όσον αφορά αρμοδιότητα τελικά επί της νομολογίας. Ωστόσο όμως ιδιαίτερα υπό το πρίσμα αυτών των πρόσφατων γεγονότων συμφωνώ ότι σε σχέση με την νομολογία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συστημική αποτελεσματικότητα διευθέτησης περιπτώσεων και καθώς επίσης και των συσσωρευτικών όρων και προϋποθέσεων η πιο εξατομικευμένων ή πιο εξειδικευμένων ε, διαδικασιών. Ωστόσο όμως αυτή θα είναι η πορεία προς τα εμπρός προς το μέλλον και ίσως ε, μπορεί να υπάρχει και κάποια αισιοδοξία ότι δηλαδή στο τέλος, τέλος δεν θα έλεγα ότι είναι το θέμα της πίεσης του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Είναι το θέμα των συνταγματικών δικαστηρίων ε, πανευρωπαϊκά και υπάρχει το θέμα του μηνύματος που αποστέλλεται από το δικαστήριο του Στρασβούργου για αυτό το ζήτημα. Διότι αυτό το οποίο έπραξε αυτή η γνωμοδότηση και είναι παράδοξο αυτό έθεσε θέματα της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο επίκεντρο. Και ίσως ε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ήταν ο κυριότερος στόχος σε σχέση με την ε, ε, γνωμοδότηση του δικαστηρίου διότι δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξουν άλλες ε, προδιαγραφές ε, για την ε, ρύθμιση αυτών των θεμάτων. Ωστόσο όμως με βάση αυτό το μήνυμα υπήρξαν πολλές αντιδράσεις συνταγματικών δικαστηρίων και από το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο αλλά και από πλευράς του Λουξεμβούργου διότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί διότι διαφορετικά ο πριτανεύων ρόλος του ευρωπαϊκού δικαίου δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να υπονομεύεται. Δεν επιθυμούσαν βέβαια το Λουξεμβούργο να έχει εκείνο αρμοδιότητες επιθεμάτων που θεωρούσαν αποκλειστική τους αρμοδιότητας. Υπάρχει τώρα ένα περιθώριο, ανοίγει η προοπτική για μια προσέγγιση μεταξύ των διαφορετικών πλευρών και αυτό μπορεί να είναι μόνο επικοδομητικό σε σχέση με το μέλλον και θα μπορέσουμε ίσως να ξεπεράσουμε, να υπερβούμε αυτά τα προβλήματα. Κύριος Ζακέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, πρέπει να πω ότι η κατάσταση που έχει προκύψει δεν είναι εντελώς δραματική όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύει ο χάρτης, εφαρμόζεται από το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και εφαρμόζεται με μια κάποια αυστηρότητα. Αυτό φαίνεται από την ομολογία του δικαστηρίου μας. Δεν βρισκόμαστε σε κατάσταση ε, νομικού κενού έλλειψης δικαίου όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Αντίθετα θεωρώ ότι όλη η κατάσταση μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να σκεφτούμε τα πράγματα. Και βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι το δικαστήριο του Λουξεμβούργου όλο και περισσότερο μέσω της ερμηνείας και μέσω της νομολογίας του συμπεριλαμβάνει πλέον τις αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μένει να δούμε απλώς αν το δικαστήριο του Λουξεμβούργου θα είναι το τελευταίο όργανο το οποίο θα ερμηνεύει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή αν θα πρέπει στη συνέχεια να προχωράμε λίγο παραπάνω και να φτάνουμε δηλαδή και στην ερμηνεία την οποία παρέχει το δικαστήριο του Στρασβούργου. Νομίζω καταρχάς ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία όσον αφορά τα επίμαχα ζητήματα. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να το πετύχουμε. Αυτό το έχουν πει πολλοί. Σαφώς υπάρχουν κάποια ουσιαστικά στη συνέχεια προβλήματα και συμφωνώ με τον κύριο Πολάκεβιτς, το ζήτημα της αμοιβαία εμπιστοσύνης πρέπει να επιληθεί, αλλά και από αυτού έχουμε σημειώσει πρόοδο. Δεν μπορούμε επί του παρόντος να δώσουμε οριστική λύση όσο δεν γνωρίζουμε την τελική νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου που ελπίζουν να την έχουμε μέσα μερικούς μήνες. Αυτή τη στιγμή θα την έχουμε, θα δούμε σε ποιο βαθμό και πού μπορούμε να πετύχουμε συνένεση και πώς μπορούμε να εργαστούμε στη συνέχεια. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να βιαζόμαστε. Νομίζω ότι μας έχει δοθεί ο παρέτος χρόνος προβληματισμού και περισυλλογής. Όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, συμφωνώ μαζί σου ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, και αναφέρομαι στον Ρικάρδο Πάσος, να έχουμε μία αναγκαστική αλλαγή των συνθήκων. Αν δούμε ότι το ζήτημα όμως δεν προχωράει, τότε ενδεχομένως θα πρέπει να καταλήξουμε και σε αυτή τη λύση. Ενδεχομένως να καταφέρουμε όμως να βρούμε μια ενδιάμεση λύση, λιγότερο ριζοσπαστική. Αυτή τη στιγμή αυτή η επιφύλαξη η οποία προτάθηκε νομίζω ότι έχει κολλήσει σε επίπεδο κρατών μελών. Από πολιτικής λοιπόν πλευράς δεν θα ήταν δικαιολογημένο και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα ήταν ιδιαίτερα σκόπιμο ισόφρον. Το πραγματικό πρόβλημα με την ΚΕΠΑ δεν έχει να κάνει με το ότι οι νομοθετικές πράξεις της ΚΕΠΑ θα μπορούσαν να παραβιάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι περισσότερες από τις πράξεις αυτές άλλωστε το γνωρίζετε, δεν είναι υποχρεωτικές. Το πρόβλημα είναι περισσότερο οι δράσεις της ΚΕΠΑ στα πλαίσια αποστολών, αποστολών με συγχωρείτε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένως στα πλαίσια αποστολών της ΚΕΠΑ να μπορούμε να έχουμε φαινόμενα κακοδιαχείρισης, φαινόμενα μη ορθή συμπεριφορά από του στρατιώτε που συμμετέχουν σε αυτέ τι αποστολέ. Εκεί πέρα τίθεται περισσότερο ζήτημα προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά όμω αποτελούν ένα τμήμα μόνο τη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι επί των, ζητημάτων αυτών θα μπορούσε να επιληφθεί το δικαστήριο του Λουξεμβούργου στα πλαίσια της ευθύνη που φέρει για την ΚΕΠΑ. Και απευθύνομαι λίγο και στο ερώτημα της κυρίας Πινέλη. Σαφώς πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε ενδεχομένω τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι ανάλογο έχουμε δει και με άλλου τομεί στο παρελθόν. Για την ΚΕΠΑ ας περιμένουμε αυτή τη στιγμή να δούμε τι θα πει το ίδιο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν χρειαστεί να ασχοληθεί με τέτοια ζητήματα. Και υπάρχει και ένα ζήτημα στρατηγικής. Αν έχουμε μια συμφωνία επί πέντε σημείων, επιστρέφουμε στο τραπέζι πραγματεύσεων πάλι με πέντε σημεία ή μήπως θα ήταν ε, καλύτερο να έχουμε μία σφαιρική τοποθέτηση και προσέγγιση θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η στρατηγική που θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι καλύτερο να επανέλθουμε με μία δέσμη προτάσεων από το να κάνουμε ξεχωριστές διαπραγματεύσεις για κάθε ξεχωριστό προβληματικό σημείο. Νομίζω ότι επ' αυτού θα πρέπει να δοθούν από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένες λύσεις. Ευχαριστώ κυρία Μωράνο. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά απόλαυσα τη συζήτηση, την επικοινωνία που είχαμε και την ανταλλαγή απόψεων. Θα σταθώ σε ένα σημείο που αναφέρθηκε πολλές φορές. Ε, το δίκαιο είναι αποτελεσματικό μόνο όταν έχει στο πλευρό του και την πολιτική βούληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υποβάλει μια καταπληκτική και ευρηματική όπως είπε κάπως προλαλή σας πρόταση ε, για να διασκεδάσει κάποιες ανησυχίες. Αν όμως δεν συνοδεύεται και από πολιτική βούληση, είναι μάταιο, γιατί σε τελική ανάλυση οι πολιτικοί ηθήνοντες αποφασίζουν και αυτοί διαμορφώνουν το δίκαιο. Οπότε, κάθε φορά ε, που έχουμε μια κρίση και το βλέπουμε από την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Είχαμε διάφορα στάδια, εξελίξεις και μετά από κάθε κρίση υπάρχει και μία νίκη. Οπότε ας μην κοιτάμε μόνο υπό αρνητικό πρίσμα τη γνωμοδότηση. Θα πρέπει να διδαχθούμε από αυτή και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε κάποια προβλήματα. Και ίσως, ε, κυρία Σπινέλη, δίκιο έχετε, ίσως ήταν ένα μήνυμα που μας έστειλε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με τη γνωμοδότηση του. Πρόσφατα είχαμε συνεντεύξεις με δικαστές ε, και οι ίδιοι ε, εξετάζουν την πιθανότητα αναθεώρηση της συνθήκης. Και η μόνη λύση που προτείναμε δεν ήταν η επιφύλαξη για την ΚΕΠΑ. Αλλά ίσως ένας τέτοιος αποκλεισμό ε, μέσω, ε, μέσω αποκλεισμός ή βράχη πρόθεσμα εξυπηρετεί. Αλλά μακροπρόθεσμα η λύση ίσως θα ήταν η αναθεώρηση των συνθήκων. Αλλά για την αναθεώρηση είναι που χρειαζόμαστε μεγάλη πολιτική βούληση. Και αυτή είναι η δυσκολία μεταξύ των δύο στοιχείων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα μπορούσε κάτι θετικό να βγει από όλα αυτά. Και επίσης πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Και η ιδέα του ψηφίσματος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν πρέπει να ε, παραμεριστεί. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το θεσμικό όργανο πολύ συχνά δίνει όθηση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή για να πραγματοποιήσουν αλλαγές. Και όλα τα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων σε αυτό το επίπεδο εξετάζονται. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολλές ευκαιρίες και πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ιδέα η ιδέα του ψηφίσματος για να προλάνει το έδαφο ε, για πιθανές αλλαγές στο μέλλον. Αυτό είναι το θετικό μήνυμα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι κάθε κρίση συνεπιφέρει και θετικές αλλαγές. Ευχαριστώ. Commission, no. Everything is in your hands. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα όπως συνήθως βρίσκονται στα χέρια σας. Πείτε και εσείς κάτι θετικό. Ευχαριστώ θερμά κυρία Πρόεδρε. Ναι, θα ήθελα και εγώ να υποβάλω κάποια σχόλια μετά από την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συζήτηση που ε, μας ενέπνευσε και εμάς και θα τα διαμηνήσω όλα και σε πολιτικό επίπεδο στους αρμοδίους. Πιστεύω ότι όλοι μας ως δικηγόροι, νομομαθείς ή πολιτικοί ε, επικρίνουμε μάλλον την γνωμοδότηση του ΔΕ που μας ευνηδίασε. Αλλά η γνωμοδότηση αυτή πια είναι ένα γεγονός και θα πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη. Και μάλιστα απορρέει από το κράτος δικαίου, γιατί το δικαστήριο του δικού μας ε, ε, νομικού συστήματος δημοσίευσε αυτή τη γνωμοδότηση. Οπότε θα πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη και να στηριχθούμε σε αυτή και στα πορίσματα του δικαστηρίου στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Σε ό,τι αφορά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Χάουρεγγι ότι ίσως ελπίζαμε σε μια ταχύτερη πρόοδο από τη γνωμοδότηση και μετά, αλλά σίγουρα έχει γίνει μεγάλη προεργασία σε τεχνικό επίπεδο. Και αισθανίζομαι πλήρως την ανάλυση του καθηγητού Ζακέ ότι για τα δύσκολα θέματα, τα πιο δυσεπίλητα, πρέπει να περιμένουμε σημαντικές αποφάσεις και των δύο δικαστηρίων που είναι απαραίτητες για τις περαιτέρω λύσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι οι αλλαγές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το απολύτως απαραίτητο για να εκπληρωθούν οι, οι προϋποθέσεις που έθεσε το δικαστήριο. Και αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να εξεταστούν και υπό το φως της μελλοντικής νομολογίας ό,τι αφορά και το εύρος της δικαιοδοσίας στην ΚΕΠΑ ή τα θέματα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων υπό το πρίσμα της αμοιβαίας αναγνώρισης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Σημείο 3 και εδώ θα διαφωνήσω με τον φίλο Ρικάρντο Πάσος γιατί κατά τη γνώμη της Επιτροπής αλλά και του Συμβουλίου καμία νέα απόφαση του Συμβουλίου που να εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαπραγμάτευση απαιτείται. Δεν χρειάζονται νέες διαπραγματευτικές οδηγίες που είναι τμήμα της απόφασης του Συμβουλίου γιατί οι διαπραγματευτικές εντολές του 2010 επαρκούν, δεν αντιβαίνουν ε, στην γνωμοδότηση του ΔΕ, τη συμπληρώνουν. Και αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να έχει διαβουλεύσει με την Ειδική Επιτροπή που συγκρότησε το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Οπότε δεν χρειάζεται νέα απόφαση για διαπραγματευτική εντόλη. Πάντως θα έχουμε διαβουλεύσει με το Συμβούλιο όσοι ήθιστε. Και μάλιστα όχι μόνο, έχουμε στενό διάλογο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέταρτο σημείο για την διαπραγματευτική στρατηγική α, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επειδή ακριβώς δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση σε πολιτικό επίπεδο, δεν μπορώ να κάνω επίσημες δηλώσεις ή δεσμεύσεις. Πάντως, συμφωνώ με τον καθηγητή Ζακέ ότι καλύτερα να έχουμε μία διαπραγματευτική θέση εφόλης της ύλης για όλα τα σημεία και μετά να επανέλθουμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Και αυτή είναι και η κρατούσα γνώμη στο Συμβούλιο ε, μεταξύ των κρατών μελών. Από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον. Και τέλος, Είναι μεν αλήθεια ότι ίσως είμαστε σε δύσκολη θέση στο Στρασβούργο, γιατί θα πρέπει να ξαναζητήσουμε επανάληψη των διαπραγματεύσεων. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει οι αλλαγέ να περιοριστούν στα απολύτω απαραίτητα, αλλά σίγουρα για κάποια σημεία θα χρειαστούν αλλαγέ στο σχέδιο συμφωνία, στην επεξηγηματική έκθεση και κάποιε διακηρύξει, δηλώσει στο διαπραγματευτικό πακέτο. για... θα πρέπει να δούμε τι θέμα θα καλυφθεί από πού και πώς. Και επανέρχομαι, επανέρχομαι στο πρώτο σημείο. Θέλουμε να υπακούσουμε και να σεβαστούμε μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το κράτος δικαίου, που είναι κοινή αξία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, μας υποχρεώνει και απαιτεί από εμά να ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση του σεβασμού, δηλαδή της γνωμοδότησης του ΔΕΕ. Επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την προσχώρηση και κάνει σχετικές διαπραγματεύσεις, όχι για να κερδίσει κάποιο πλεονέκτημα οικονομικό ή πολιτικό για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για ενταχθεί σε αυτό το πανευρωπαϊκό σύστημα της προάσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οπότε η κατάσταση είναι αυτή εξ αρχή πολύ διαφορετική από ότι η κατάσταση σε άλλε διεθνεί διαπραγματεύσει. Και νομίζω ότι αυτή είναι η κοινή αντίληψη και ημών και του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Φτάνουμε στο τέλος της συζήτησής μας. Ξέρετε ότι ε, η δημόσια αυτή ακρόαση μεταδίδεται και μέσω του διαδικτύου. Καταγράφουμε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Συντοποιούμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια πρόκληση όσον αφορά το όλο χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Νομίζω πάντως ότι ε, θα πρέπει να μας ασκηθεί και κάποια πίεση, αν θέλετε, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα αυτό, γιατί άλλωστε προβλέπεται η υποχρέωση της τελικής προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ούτως ή άλλως. Αλλά υπάρχει και ένας επίγον χαρακτήρας όσον αφορά τις πολιτικές ανάγκες, την πολιτική πτυχή του ζητήματος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πολλές αλλαγές, πολλές προκλήσεις, γινόμαστε και εμείς όλο πιο ευαίσθητοι και δεκτικοί για τα ζητήματα αυτά που σχετίζονται με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν το ζήτημα αυτό πολύ σημαντικό και από πολιτικής πλευράς. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των επιτροπών μας να συμβάλλουμε κι εμείς και να υποστηρίξουμε την όλη διαδικασία ολοκλήρωσης της προσχώρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ. Προφανώς θα πρέπει να δούμε και πώς εξελίσσεται η νομολογία και στα δύο δικαστήρια και αυτό θα μας εμπνεύσει και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ βέβαια στο να ολοκληρώσετε την προσχώρηση Μία ελπίδα που τρέφουμε από τη δική μας την πλευρά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι ελπίζουμε ότι ακόμα και αν το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, δεν θεωρήσει ότι θα πρέπει να δοθεί νέα διαπραγματευτική εντολή, εσείς στα πλαίσια της εφιστάμενης διαπραγματευτική εντολή θα καταφέρετε να καταλήξετε τελικά σε μια συμβαστική λύση, έτσι δεν είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθο, δίστανται ελαφρώ οι απόψει ανάμεσα στα δύο όργανα όσον αφορά τη διαπραγματευτική εντολή. Θεωρώ ότι και στα πλαίσια τη υφιστάμενη διαπραγματευτική εντολή, εφόσον δεν ενωθεί θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Μιλώ εκπρόσωπο Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ναι, μα προφανώ. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπώντα την Ευρωπαϊκή Ένωση, ολοκληρώσει τη δέσμη προτάσεων, εμεί θα ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει. Είναι το μόνο που περιμένουμε άλλωστε εμεί στο Στρασβούργο. Άλλωστε, α μην ξεχνάμε ότι μία προτεραιότητα πρωταρχική σημασία για το Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες που εκπροσωπούνται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και που εν τέλει θα αποφεληθούν από την όλη διαδικασία είναι να τροποποιηθεί η υφιστάμενη εκκρεμής κατάσταση. Γιατί αυτή τη στιγμή η ε, υφιστάμενη αυτή κατάσταση δημιουργεί πάρα πολλές αμφισημίες και για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και για τους ίδιους Ευρωπαίους πολίτες. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή σας. Αναφέρομαι σε όλους τους προσκεκλημένους και νομίζω ότι ε, σε οτιδήποτε και να καταλήξετε θα ήθελα πραγματικά να ενημερώνετε παράλληλα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ή κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων ή κατά την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων. Ολοκληρώνεται λοιπόν το σημείο αυτό. Ας κάνουμε ένα 15 λεπτό διάλειμμα και ας συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα σημεία της ημερήσιας διάταξης στις 11.30. 15 λεπτό λοιπόν διάλειμμα. <laughs> Συνάδελφοι, συνεχίζουμε παρακαλώ με το επόμενο σημείο που είναι η δημοσιονομική ικανότητα στην Ευρωζώνη, συνέπειες για τον προπολογισμό, συμπληρωματικότητα και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δυνάμει του άρθρου 54 αναθέσαμε την έκθεση στον Παύλο Ρανζέλ. Αν θέλει να μιλήσει, να περάσουμε κατευθείαν στους και Paolo, σε ακούμε. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, όπως ξέρετε, εκπονούμε γνωμοδότηση για το θέμα της δημοσιονομικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως πρώτο θέμα θα ήθελα να πω ότι ως συνήθως, οι γνωμοδοτήσεις μας πρέπει να είναι πολύ σύντομες. Έχουμε συγκεκριμένο αριθμό στοιχείων. Πολύ περιορισμένο, πολύ μικρό και δεν μπορούμε να καλύψουμε αυτά τα περίπλοκα θέματα. Τούτου λεχθέντος ε, να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για μία προσωρινή εκδοχή έγινε αναβολή από την Αρμόδια Επιτροπή και μια και έχουμε χρόνο μέχρι την οριστική εκδοχή μπορούμε να έχουμε την εξέταση σήμερα. Ήδη συναντήθηκα με τους ε, συνεισηγητές Μπέρες και Μπέγκε από τις Επιτροπές Προϋπολογισμών και ΕΚΟΝ και έχουμε καλά γραφά, αλλά παρά είναι ανοιχτά. Δεν ξέρουμε αν θέλουμε μια δημοσιονομική ικανότητα που θα προσανατολίζεται στην απορρόφηση των ασύμετρων κραδασμών ή σε συστήματα ασφάλισης κατά της ανεργίας ή σε μηχανισμούς σύγκλησης ε, ή αλληλεγγύης και πλέον υποστήριξη για τη χρήση των διαφορετικών ταμείων. Οπότε δεν ξέρουμε τι εννοούν με την περιορισμένη δημοσιονομική ικανότητα. Πάντως, ε, για μας στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να αναπτύξουμε πλήρη δημοσιονομική ικανότητα στην Ευρωζώνη. Κάτι που θα ήταν ευκταίο, αλλά κάτι τέτοιο προϋποθέτει αναθεώρηση των συνθήκων. Χρειαζόμαστε αλλαγή των συνθήκων για να φτάσουμε σε πλήρη δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Βέβαια υπάρχει κάποιο περιθώριο ε, από συνταγματική άποψη και δεδομένα των συνθήκων για μια περιορισμένη έστω δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Και αυτό είναι απαραίτητο απολύτως απαραίτητο για να συμπληρώσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η οικονομική διακυβέρνηση δεν νοείται χωρίς έστω και μια περιορισμένη δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι σαφές και στο, στην έκθεση των πέντε πρόεδρων. Βέβαια και η έκθεση αυτή ε, προβλέπει αναθεώρηση των συνθήκων αλλά προς το παρόν δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει αρκετό περιθώριο. Ε, δεν ασχολούμαστε καν με την αναθεώρηση των συνθηκών. Επικεντρωνόμαστε σε πιο βραχυπρόθεσμες ε, ενέργειες με βάση το ισχύον θεσμικό και συνταγματικό πλαίσιο. Τι μπορούμε να πούμε τώρα για το θέμα αυτό. Θα μπορούσε να γίνει στα πλαίσια του κοινοτικού προπολογισμού, που είναι η συνέπεια της αρχής της ενότητας του ενιαίου χαρακτήρα του προπολογισμού, που κατοχυρώνεται στις συνθήκες και αναφέρεται και από τους συζητητές. Η ενότητα του προπολογισμού. Και φυσικά ε, με σεβασμό των αιτήσεων πολιτών, ε, των δημοσιονομικών ε, πλαισίων. Μπορούμε να αυξήσουμε το ανώτατο όριο ιδίων πόρων, να προβλέψουμε νέες κατηγορίες ιδίων πόρων, ακόμη και αν προέρχονται από ορισμένα κράτη-μέλη. Και μπορούμε επίσης να προβλέψουμε ένα εισόδημα για να χρηματοδοτήσουμε ειδικέ δαπάνες. Για παράδειγμα, ένα σύστημα ασφάλισης ε, κατά της ενέργειας. Αν αυτό τελικά ε, περιλάβει στην έκθεσή της Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Ε, οι συνθήκε προβλέπουν κάποιε εγγυήσει για τον ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό για συγκεκριμένε επιχειρήσει επιχειρήσεις ε, και ε, στα πλαίσια του κανονισμού του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου έχουμε ιδιαίτερου ειδικού μηχανισμούς που προβλέπουν κινητο, κινητοποίηση των κονδυλίων πέραν των του προϋπολογισμού και των των ορίων, όπως είναι το EFCM και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Το θέμα δεν είναι να έχουμε επικάλυψη συστηματική υπέρβαση των ανωτάτων ορίων, αλλά απλώ υπάρχει δυνατότητα να ξεπεράσουμε τα, τα ανώτατα όρια. Αυτό το προβλέπει ο ίδιος κανονισμός του Πουδουπού. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα υπέρβασης ως δημοσιονομική ικανότητα. Δηλαδή δεν θεσπίζουμε νέα εξαίρεση, απλώς χρησιμοποιούμε αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε το, παράδειγμα του EFSEM ή του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση που επιτρέπουν την υπέρβαση των ανώτατων ορίων. Μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις επιτρέπεται τέτοιου είδους ικανότητα. Αυτή είναι η θεσμική προσέγγιση σε αυτό το μηχανισμό μπορεί όμως να αλλάξει, να τροποποιηθεί στην τελική διατύπωση. Στο τέλος θα έχουμε τότε ένα ακριβέστατο όραμα επισκόπηση του τι προτείνεται από τους εισηγητές της ΕΚΟΝ. Και έτσι θα υπάρξουν αυτές οι αλλαγές. Υφίστανται όμως πραγματικά συνταγματικά ζητήματα, θέματα συμβατότητας με τη συνθήκη και θα πρέπει να τα επισκοπήσουμε και να αναθεωρηθούν διότι είναι ανοιχτή διαδικασία και το πλαίσιο αυτό και οι διαδικασίες από πλευράς εισηγητών και δεν μπορέσαμε αυτό το θέμα να το διευθετήσουμε με απολυτότητα. Δεν είμαστε βέβαιοι δηλαδή ποια θα είναι η τελική επιλογή και διατύπωση των εισηγητών. Σε αυτή τη φάση όμως μπορούμε με σαφήνεια να πούμε ότι πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό το πλαίσιο. Πρώτον, υπάρχει ανάγκη νομιμοποίησης δημοκρατικής ε, όσον αφορά και τον έλεγχο από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δημοσιονομική ικανότητα και δυνατότητα που πραγματικά εμείς ε, σε αυτήν προσβλέπουμε θα έπρεπε φυσικά να ελέγχεται ως διαδικασία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να εντάσσεται στην διαδικασία λήψης ε, δημοκρατικών αποφάσεων με την ε, εμπλοκή του Ευρωκοινοβουλίου πάντα συνάδοντας με τη συνθήκη, ευθυγραμμιζόμενη με τη συνθήκη. Εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα, ίσως και συνταγματικής ε, υφής. Αν δεν είχαμε μια τέτοια αρμοδιότητα θα περιοριζόμαστε μόνο στην Ευρωζώνη. Πρέπει να σχεδιάσουμε την εμπλοκή μας με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την ε, ιδιότητά μας αυτή και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Αρκετά υπάρχουν για να εκπονηθούν και αυτό θα σημαίνει μια νέα έκθεση μετά την έκθεση ΕΚΟΝ, αν αυτή και όταν εγκριθεί εκείνη για την ανάπτυξη του δικού μας δυναμικού. Πώς μπορεί αυτό δηλαδή να εκπονηθεί και να λειτουργήσει. Και πιστεύω ότι αυτό δεν θα εντάσσεται στην ίδια τη δική μας γνωμοδότηση. Όμως έχουμε μια φιλοδοξία που μας εμπνέει. Δηλαδή την λύση που είχε προταθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό Τραπεζών. Όπως γνωρίζετε αυτό το συζητήσαμε όταν συντάξαμε την έκθεσή μας ε, για την έκθεση για την έγκριση εποπτικών λειτουργιών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε μια συζήτηση, θα ήταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μέχρι ποιου βαθμού. Όταν ε, αποφασίστηκε ότι θα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όταν συμφωνήθηκε αυτό και ε, σε σχέση με τις επιλογές του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φυσικά υπήρξε έγκριση διότι κάποιες χώρες που ήταν υποψήφιες χώρες ε, για να ενταχθούν στο ευρώ όχι εκείνες που έχουν το opt-out την αυτοεξαίρεση αλλά εκείνες που έχουν αναλάβει την υποχρέωση να ενταχθούν στο ευρώ κάποιες επιτράπει να συμμετάσχουν αν επιθυμούν στην εποπτεία αυτήν όσον αφορά την έκτο ε, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι υπάρχουν συγκεκριμένα πλέον σε σχέση με την εφοπτεία. Και έτσι φυσικά θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή τους στο Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο γι' αυτό. Σύμφωνα με τις συνθήκες λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει τον τελευταίο λόγο και σχεδιάσαμε ένα μηχανισμό όπου το σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα λαμβάνει απόφαση και θα εγκρίνεται από το σώμα των 19 ε, συμμετεχόντων μελών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει με, γνωμοδοτη... Ε, επιχειρηματολογημένη γνωμοδότηση να ε, αναφέρεται σε αυτό. Οι, μη, ε, οι χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη μπορούν λοιπόν να λάβουν μια τέτοια απόφαση. Στο τέλος, τέλος όμως αυτό μπορεί να είναι σπάνιο, παρότι μπορεί να συμβεί, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να είναι διαφορετική από το, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόκειται για κάτι δηλαδή στο οποίο δεν, έχουν, δεν έχει υπάρξει ακόμα συμμετοχή. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένα κίνητρο λοιπόν στις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη να κινητοποιηθούν και να ενταχθούν στην Ευρωζώνη. Αν έχουν όλα τα προτερήματα της Ευρωζώνης και μπορούν ε, να έχουν το δικό τους νόμισμα, αυτό δεν επιλύεται. Πρέπει λοιπόν ε, για όλους αυτούς τους λόγους να ε, δημιουργηθεί ένα τέτοιο περίπλοκο σύστημα. Δεν λέω ότι πρέπει να επαναληφθεί η υιοθέτηση αυτής της λύσης, λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια λύση που θα διασφαλίζει ότι οι χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη σε σχέση με αποφάσεις που έχουν επιπτώσεις άμεσα στις χώρες Ευρωζώνης αν θέλουν να ενταχθούν σε, αυτή την, σε αυτό το δυναμικό αν θέλουν να είναι παρούσες αυτές οι χώρες μπορούν να έχουν ένα λόγο που θα αρθρώνουν και σε σχέση με τις ε, επιπτώσεις που θα υπάρχουν για την ε, ζώνη ε, του ευρώ θα πρέπει να συμμετέχουν τα κράτη της ζώνης αυτής ώστε οι επιπτώσεις να είναι δεδομένες στο εύθετο πλαίσιο. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο δεν είναι καθόλου τόσο εύκολο να αντιμετωπιστεί δεν είναι τόσο εύκολο να επιλύθει και είναι το θέμα της εμπλοκής των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών. Φυσικά το να υπάρχει περιθώριο να εμπλακούν υπό το πλαίσιο των πρωτοκόλων είναι κάτι δεδομένο και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως ε, επιλογή, ως εναλλακτική λύση όμως φυσικά πάντα σεβόμενοι τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας ε, υπάρχει πάντα και μια τύπη συνεργασία που ε, είναι δεδομένη. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να επιτευχθεί ο έλεγχος ε, των ευρωπαϊκών αποφάσεων από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα Εθνικά Κοινοβουλία θα ελέγχουν τις εθνικές κυβερνήσεις και ιδιαίτερα τη συμμετοχή των εθνικών κυβερνήσεών τους στο Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ελέγχει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια ενδεχόμενα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αν δημιουργήσουμε ακριβώς και ένα ε, σώμα, ένα διοικητικό συμβούλιο για την ε, ε, δυνατότητα, την ικανότητα αυτή πρέπει να υπάρχει και ένα σώμα για την ελεγκτική δραστηριότητα. Τώρα, ο έλεγχος θα πρέπει να παραμένει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να διαφοροποιούμε αυτά τα ζητήματα. Αυτό θα πρέπει να είναι το κύριο θέμα που θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν υπάρχει απόλυτα επαρκές περιθώριο για να αναπτυχθούν όλα αυτά. Εδώ πρέπει οι αρχές να αναπτυχθούν αρχή κοινοβουλευτικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αρχή της εμπλοκής των Εθνικών Κοινοβουλίων υπό τα ενισχύει πρωτόκολλα και φυσικά η συμμετοχή της, η δυνατότητα συμμετοχής των χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη με έναν τρόπο ώστε τουλάχιστον να μπορεί να διασφαλίζεται η συμμετοχή τους αυτών των χωρών αλλά όχι με το ίδιο καθεστώς σε σχέση με τις χώρες που ανήκουν οι ίδιες αυθεντικά στην Ευρωζώνη. Αυτό θα είναι κάπως δύσκολο και ευαίσθητο να μπορέσει να διευθετηθεί μέσα στο πλαίσιο των, ε, ε, της παρούσας διοργάνωσης που υφίσταται συνταγματικά εδώ και από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όμως μπορεί να είναι εφικτό και δυνατό αυτό αν υπάρξουν, μια τέτοι, αν υπάρξουν τέτοιες προοπτικές θα μπορέσουν πιο εύκολα να διευθετηθούν και να σχεδιαστούν λύσεις. Αλλά είναι φυσικά τόσο δύσκολο να τροποποιηθούν οι συνθήκες ώστε ίσως ε, μια τέτοια λύση δεν θα είναι πιθανή θα έλεγα πρόθεσμα. Είμαι στη διάθεσή σας για παρατηρήσεις και σχόλια και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε. Δεν θέλω όμω μόνο κάποιε παρατηρήσεις, δεν θέλω να σα ανησυχήσω. Είναι οι σκιώδεις ηγητέ αυτοί οι οποίοι θα μιλήσουν και καταρχάς η κυρία Μπρεσό εξ ονόματο των σοσιαλιστών. Καταρχάς, σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον Πάουλο Ράντζελ. Δεν πρόλεβα να διαβάσω παρά μόνο πάρα πολύ γρήγορα το κείμενο αυτό, το έγγραφο εργασία γιατί το λάβαμε την τελευταία στιγμή και ενώ συζητούσαμε τελικά για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα το πρωί το έλαβα το έγγραφο αυτό λοιπόν. Πάντως τόσα μόλις τώρα μας είπες μου φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα. Αυτό το οποίο βλέπω στην πράξη είναι ότι Πολλά πράγματα ακόμα πρέπει να μας απασχολήσουν, ιδίως όσον αφορά τη θεσμική συνταγματική πτυχή του ζητήματος και πιο συγκεκριμένα πως αυτά μπορούν να συνδυαστούν με την πρόταση για μια δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Αν κατάλαβα καλά τα όσα μας είπες, Νομίζω ότι μας δίνεται τώρα δυνατότητα στα πλαίσια των συνθήκων να δημιουργήσουμε μια δημοσιονομική ικανότητα για την Ευρωζώνη. Εσύ μας είπες ότι μπορεί να μην είναι τόσο ευρύ αυτή η δημοσιονομική ικανότητα. Το θέμα δεν είναι τόσο το εύρος, το θέμα δεν είναι ποσοτικό, το θέμα είναι τα μέσα τα οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα ιδίων πόρων που θα μας επιτρέψει τελικά να έχουμε μια δημοσιονομική ικανότητα για την Ευρωζώνη. Και κατά αυτόν τον τρόπο και στην έκθεση Μπροκ το βλέπουμε αυτό, μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον ένα τμήμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού το οποίο θα δίδεται για την Ευρωζώνη. Και αυτό πάλι στα πλαίσια του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά θα αποτελεί σίγουρα προϋπολογισμό πλέον για την Ευρωζώνη. Ένας προπολογισμό αφιερωμένος στην Ευρωζώνη. Ως Επιτροπή λοιπόν Σταγματικών Υποθέσεων και μέσω συγκεκριμένων τροπολογιών θα μπορούσαμε να δούμε ποια θα είναι η μέγιστη αυτή διάσταση, αν θέλετε, που μας δίνεται για τη δημοσιονομική ικανότητα στα πλαίσια των συνθήκων τι εύρο που θα είναι το πεδίο εφαρμογή δηλαδή αυτή της δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Πρέπει βέβαια πρώτα να δούμε και την ίδια την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, τι τελική μορφή θα πάρει δηλαδή. Δικό μας καθήκον θεωρώ στα πλαίσια της δικής μας Επιτροπής είναι να οριοθετήσουμε το εύρο λειτουργία αυτή τη δημοσιονομική ικανότητα της Ενδεχομένως να μπορούσαμε και μέσω τροπολογιών να διευρύνουμε και την ίδια την έκταση του, της γνωμοδότησής σου, γιατί ξέρεις ότι μέσω τροπολογιών μπορούμε να προσθέσουμε περισσότερα στοιχεία. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή μέσω των τροπολογιών να συνδυάσουμε τις διαφορετικές απόψεις και θα προσπαθήσουμε βέβαια από τη μία έκθεση στην άλλη να υπάρχει και ένα υψηλό επίπεδο συνεκτικότητας και συνοχής. Το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια ενιαία κοινή θέση ως Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μέσσερος από τους συντηρητικού μεταρρυθμιστές. Φαντάζομαι δεν θα εκπλήξει τον καταπληκτικό μας ηγητή ότι η ομάδα μας δύσκολα θα υποστηρίξει την γνωμοδότησή σας κύριε Ραντζέλ. Περισσότερο όμως για θέματα αρχής. Α, ταμείο Παγκοσμιοποίησης, ήδη έχουμε διαφωνίες επί της αρχής. Πέραν των αντίρρησεων όμως, να κάνω κάποια σχόλια. Καταρχήν ως προς την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σημαντικό θέμα. Ο εισηγητής μας είπε ότι και για τον ίδιο είναι σημαντικό να υπόκειται η έκταση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εγώ δεν συμφωνώ. Α, καλά. Να συμφωνούμε. Αν συμφωνούμε ακόμη καλύτερα, γιατί η ανεξαρτησία της έκτη είναι προφανώς σημαντική. Απ' την άλλη, με ικανοποίησαν τα σχόλιά σας για τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μακάρι να συμφωνήσουμε να διευρυνθεί ο έλεγχος αυτός, όχι μόνο ε, έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ε, συλλογικό όργανο, αλλά και έλεγχος επί των μεμονωμένων επιτρόπων. Στο σημείο 4 ο εισηγητή μας υπενθυμίζει ότι η ικανότητα αυτή θα πρέπει να αποτελεί θέμα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα μένει να αποφασιστεί. Αν η Βρετανοί μας ψηφίσουν ναι στο δημοψήφισμα, τι θα γίνει. Υπό αυτές τις συνθήκες το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να πληρώνει για να διασώζονται ή να συμβάλλει οποιοδήποτε, οποιοδήποτε τρόπο για, να, για τις χώρες Ευρωζώνης. Και επίσης, αν χρησιμοποιηθεί γι' αυτό ο, κοινός, ο κοινοτικός προϋπολογισμός, θα πρέπει να δοθεί ένα αντιστάθμισμα, ένα αντίβαρο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα ήταν καλύτερο να θεσπιστεί ξεχωριστός προϋπολογισμός της Ευρωζώνης και όχι να εντάσσεται αυτός στον γενικό προϋπολογισμό ή τουλάχιστον, τουλάχιστον, δεν ξέρω τελικά πότε θα ψηφίσουμε, αλλά ε, να περιμένουμε για να δούμε τι τύχη θα έχει η Συμφωνία Κάμερον με τα θεσμικά όργανα και αν εφαρμοστεί, που κατά τη γνώμη μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Η Σιλβί Γκουλάρ από τους Φιλελεύθερους, σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή μας τον κύριο Ραζέλ. Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και χαίρομαι που ασχολούμαστε στην Επιτροπή μας γιατί βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Όπως ακούσαμε, το Βρετανικό δημοψήφισμα θα σκίσει μεγάλη επιρροή. Αλλά την απόφαση μας θα πρέπει να την πάρουμε εξάρτητα από αυτό. Έχουμε δύο πιθανές επιλογές. Ή θα ψηφίσουν ναι οι Βρετανοί. Αντί ε, αυτή την ο συγκεχημένο και αφήσιμο χαρακτήρα αυτή τη διεθνού συμφωνία που κανένα δεν ξέρει με ακρίβεια τι ισχύ έχει, από ό,τι ξέρω δεν θα υποβληθεί σε κύρωση στις εθνικές βουλές, οπότε τελούμε πλήρη συγχύση. Τι θα γίνει αν τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία. Γιατί αυτή η συμφωνία θεωρητικά θέτει τέρμα σε μία αρχή της συνθήκης του Μάστριχτ, ε, στο ενιαίο νόμισμα με ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Γιατί Με βάση το ότι κάποιοι ε, κάποιες χώρες ε, είχαν, θα είχαν λόγο και δεν ε, συμμετείχαν στο νόμισμα. Βέβαια, ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι αν ψηφίσουν ναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συζήτηση θα, μετατρα... θα μετατεθεί σε άλλα κρατημέλη. Και η έλλειψη δημοκρατικής διαδικασίας στην συμφωνία αυτή, γιατί έχει παρακαμφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και η έλλειψη ανάμειξη των Εθνικών Κοινοβουλίων κάνει όλα αυτά τα πράγματα κάπω αβέβαια. Και τι θα γίνει και πώς θα επηρεάσει η έκβαση του ψηφίσματο όλα αυτά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το προσδιορίσουμε αυτό στην Ευρωζώνη με τις παρούσες και μελλοντικές χώρες και υπάρχουν μακροοικονομικοί λόγοι, λόγοι λογοδοσίας που μας αναγκάζουν να προχωρήσουμε σε ένα ξεχωριστό προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Και χαιρετίζω το έργο και της συζητήτριας ε, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, γιατί είναι πραγματικά πολύ μεστή η έκθεσή της ε, και περιεκτική. Τώρα, μερικές αρχές ε, που θα ήθελα να κατοχυρώνουμε στη δική μας γνωμοδότηση. Ε, καταρχήν, να, να λέμε ότι υπάρχουν δικαιώματα που συνοδεύονται από υποχρεώσει. Δεν θα πρέπει να έχουμε ένα θεσμικό σύστημα που άνθρωποι που δεν συμμετέχουν σε ε, μία ζώνη να έχουν λόγο σε αυτήν. Όσοι συμμετέχουν θα πληρώνουν και θα έχουν λόγο και όσοι βρίσκονται εκτός ούτε θα συμμετέχουν και ούτε θα έχουν δικαιώματα που υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις τους. Μία αντιστοιχία λοιπόν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων γιατί έχουν βαρεθεί οι πολίτες μας περίπλοκες δομές και μορφώματα που δεν καταλαβαίνουν. Επίσης χαίρομαι που στο έγγραφο της ΕΚΟΝ αναφέρονται οι επιμέρους λειτουργίες του προπολογισμού. Θα ήταν επικίνδυνο να περιοριστούμε μόνο σε προϋπολογισμό που έχει μια συγκεκριμένη ε, λειτουργία. Έχουμε το θέμα του δημόσιου αγαθού, έχουμε τη λειτουργία την αντικυκλική, έχουμε την λειτουργία ανακατονομής. Θα πρέπει να τολμήσουμε να τα αναφέρουμε όλα αυτά. Γιατί τα χρειαζόμαστε. Επίσης, αυτό που είπε ο συγκητής για τα εθνικά κοινοβούλια, που και αυτά έχουν ρόλο γιατί ήμουν εισηγήτρια στο εξάπτυχο ε, σχέδιο, την εξάπτυχη πρόταση που τάχθηκε υπέρ της ανάμειξης του των Εθνικών Κοινοβουλίων. Γιατί αν μπερδέψουμε τα επίπεδα ευθύνη και αρμοδιοτήτων, θα έχουμε μια κατάσταση όπου σε τελική ανάλυση δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε λογοδοσία από τους αρμοδίους. Το θέμα της λογοδοσίας του ΕΚΤ νομίζω ότι είναι κάπως εκτός θέματος, γιατί το θέμα είναι η ε, δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Δεν είναι αυτό το θέμα της ΕΚΤ, ούτε η ΕΚΤ θα διαχειριστεί αυτή τη δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Ε, λεπτό θέμα, αλλά εκτός θέματος το θέμα της ΕΚΤ. Πάντως ε, θα ήθελα να παροτρύνω τον κύριο Ραζέλ να είναι φιλόδοξος και να μην παρασυρθεί από τους απεσιόδοξους που κρίνουν τα αιτήματα αυτά ουτοπικά. Γιατί αν ε, ξεχάσουμε τις ανάγκες του κόσμου θα μείνουμε σε μια κατάσταση κενό και θα δυσαρεστήσουμε τους συμπολίτε μας. Ευχαριστώ. Ο Χέλμουτ Σόλτς αποσιάζει και ο Φάμπιο Καστάλντο το ίδιο. Οπότε δεν έχουμε άλλους εκπροσώπους από τις πολιτικές ομάδες, άλλους και όδης Παίρνουμε στη γενική συζήτηση, ο Γιολάινα. Μάλιστα, ευχαριστώ κυρίως τον εισηγητή μας Παύλο Ρανζέρ. Η γνωμοδότησή μας πρέπει να είναι σύντομη βέβαια. Και νομίζω τα ουσιοδέστερα σημεία τα ανέφερε σωστά εκείνα τα οποία μας αφορούν ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αυτά ξεκινούν με την αναγκαιότητα της δημοσιονομικής ικανότητας για την Ευρωζώνη η οικονομική κρίση μας δίδαξε ότι η νομισματική ένωση έχει τεράστιες ελλείψεις. Στέκεται σε ένα πόδι μόνο. Το δεύτερο πόδι με την οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα απουσιάζει, δεν την έχει αυτήν. Αναγνωρίζεται ότι πρέπει να υπάρξει η δημοσιονομική ικανότητα βέβαια και θα υπέρθει Εμείς από πλευράς Ευρωκοινοβουλίου είπαμε, λέγαμε πάντα ότι πρέπει να εντάσσεται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αυτή θα ήταν η πρώτη μας επιλογή ως εναλλακτική λύση. Διότι τότε το δικό μας το Κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο θα ασκεί τον έλεγχο. Πρέπει να είμαστε κατά μιας ημι διακυβερνητικής ή καθαρά διακυβερνητικής δομής που πάλι θα μας δυσχέρεναν το βίο και πάλι θα μας άφηναν στο περιθώριο εκτός, εκτός δηλαδή αρμοδιοτήτων όσον αφορά τα δικαιώματά μας. Εμείς γενικά δηλαδή λέμε ότι η δημοσιονομική ικανότητα πρέπει να εντάσσεται ως τμήμα του προϋπολογισμού στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Γνωρίζω από τους συναδέλφους της ΕΚΟΝ, της ε, Οικονομικής Νομισματικής Επιτροπής, υπάρχουν κάποια ερωτήματα και προβλήματα για το πώς δηλαδή θα επιτευχθεί αυτό. Όμως δίνει την δυνατότητα αυτή η συνθήκη. Η συνθήκη της Λισαβόνας προσφέρει αυτή τη διαφοροποίηση ως ικανότητα, ως δυνατότητα και στο πρωτογενές δίκαιο υπάρχει η δυνατότητα ένας ειδικό προϋπολογισμός να εντάσσεται στον γενικό προϋπολογισμό. Τώρα δεν πρόκειται για μεγάλες ε, μίζωνες ε, διαπραγματεύσεις για το περί πρόκειται εδώ όσον αφορά την δημοσιονομική ικανότητα. Αυτό σίγουρα θα το διευθετήσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Νομισματικών Υποθέσεων. Όσον αφορά την μη σώροπη σχέση δηλαδή στην Ευρωζώνη θα πρέπει να υπάρξει αντιστάθμιση, θα κοστίσει αυτό και δεύτερον η δημοσιονομική ικανότητα αν μπορεί να το επιτύχει αυτό, αυτό φυσικά απαιτεί μια τελείως διαφορετική βάση για τη συζήτηση για τις μεταφορές κονδυλίων, financial transfers και τα συναφή. Εδώ φυσικά τους κραδασμούς που μπορεί να υποστεί μια χώρα ε, πρέπει να τους δούμε καθώς επίσης ε, και την ανάγκη προσαρμογών ώστε δηλαδή να μην απεμπολίσουμε δικές μας ε, αρμοδιότητες και δικαιώματα όσον αφορά το νόμισμα. Οι προσαρμογές που πρέπει να γίνουν είναι πρόδειλες, είναι προφανείς και οι διαφορετικές ε, τροποποιήσεις και μεταρρυθμίσεις και αλλαγές πρέπει να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Τώρα θα τοποθετηθούμε για το ποιος θα είναι υπεύθυνο για αυτή την δημοσιονομική ικανότητα. Ένα ταμείο, ένας ταμείας ή ένας υπουργός οικονομικών ή ένας αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως αυτό θα μπορούσε να ήταν η λογική συνέπεια των πραγμάτων αν αυτά όλα ενταχθούν στην, ε, στον Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια εποπτεύουσα αρχή, ένα είδος ταμείο, ή, ταμείου ή ένα είδος εποπτικής αρχής από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διορθώνει ο μιλητής. Ναι. Και Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ποιο ρόλο θα διαδραματίζει σε σχέση με όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο δικό μου πρότυπο που επιλέγω εγώ δεν, έχει τέτοι, δεν θα είχε τέτοιες αρμοδιότητες, θα βρισκόταν στο περιθώριο. Τον ρόλο θα αναλάμβανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και σίγουρα και το Συμβούλιο, δηλαδή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τώρα, ενδιαφέρον αρχίζει να γίνεται το θέμα όσον αφορά τη δημοσιονομική ικανότητα για την Ευρωζώνη σε σχέση με εκείνες τις χώρες που δεν είναι ακόμα μέλη της Ευρωζώνης. Και εδώ τίθενται ερωτηματικά που πρέπει να απαντηθούν. Και πάλι επαναλαμβάνω, θα εξαρτηθεί από το πού θα προέλθουν αυτά τα κονδύλια. Αν θα προέρχονται αυτά τα κονδύλια από χώρες της Ευρωζώνης, για παράδειγμα, ε, τότε φυσικά σε πρώτο λόγο οι χώρες της, Ευρωπαϊκής, ε, της Ευρωζώνης θα πρέπει να υποφελούνται από το εγχείρημα. Αλλά φυσικά για τις χώρες που θα ενταχθούν μελλοντικά στην Ευρωζώνη πρέπει να προβλέψουμε τις διαδικασίες προσαρμογής ε, απόσβεση των κραδασμών όταν θα ενταχθούν στην Ευρωζώνη. Άλλο τελείως διαφορετικό πρόβλημα είναι η, Ευρω... η Μεγάλη Βρετανία. Βρίσκεται στο περιθώριο αυτών των πραγμάτων. Ελπίζουμε βέβαια η Μεγάλη Βρετανία να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργούνται ζητήματα επειδή υπάρχουν πολλά τομείς που δημιουργούν κάποια διαφάνεια. Όμως ε, είναι σαφές ε, ότι η Μεγάλη Βρετανία η ίδια θα πρέπει να θελήσει να ενταχθεί περισσότερο στην Ευρωζώνη και ότι δεν θα υπάρχει δικαίωμα αρνησή κυρίας ε, στις περαιτέρω εξελίξεις της Ευρωζώνης από πλευράς Μεγάλης Βρετανίας. Αν θυμηθούμε τα θέματα αυτά σε σχέση με τις μεταφορές κονδυλίων και σε σχέση με το που, από πού θα προέλθουν αυτά τα κονδύλια σε σχέση με τις χώρες της Ευρωζώνης ή τις χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωζώνης δεν κατανοώ γιατί θα πρέπει να αντισταθμιστούν αυτά τα ζητήματα με πρόσθετα κονδύλια που θα καταβάλλονται στην ε, Μεγάλη Βρετανία. Να βρεθεί δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία και σε μια δεύτερη τροχιά απαιτήσεων για αντισταθμίσεις ε, και επιστροφές. Τίθενται λοιπόν αυτά τα ερωτήματα στον που πρέπει να απαντήσει. Είναι ερωτήματα αρκετά δύσκολα στην απάντησή τους. Ευχαριστώ κυρία Μπερές παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ και παίρνω το λόγο εδώ ως συνεισηγήτρια της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και Νομισματικής Πολιτικής. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον Πάολο Ραντζέλ για το σχέδιο αυτό γνωμοδότησης. Πρώτη φορά βλέπουμε ένα προσχέδιο μάλλον γνωμοδότησης, καινοτόμε προσέγγιση. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το έγγραφο εργασίας κάποια πρώτα στοιχεία, κάποιες πρώτες δυσκολίες που προκύπτουν από το ζήτημα αυτό που πιστεύω ότι θα καταφέρουμε όμως να επιλύσουμε. Και νομίζω ότι και η δική σας η Επιτροπή θα καταφέρει να συμβάλλει μέσω της γνωμοδότησής της στην εκπόνηση της τελικής μας έκθεσης. Ξέρω ότι η δική σας ε, η Επιτροπή θέλει να πετύχει την κατάλληλη θεσμική και σταγματική ισορροπία σε σχέση με το μήνυμα το οποίο θέλει να περάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή οποιοδήποτε και είναι το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα στον Ηνωμένο Βασίλειο οποιοδήποτε και αν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο αυτού τίθεται το ζήτημα της λειτουργίας τη Ευρωζώνης. Έχουμε επίσης την έκθεση Μπρεσό, έχουμε και την έκθεση Φερχόφστατ που θα ακολουθήσουν στο άμεσο μελλοντικό διάστημα και οι τρει λοιπόν αυτές εκθέσεις νομίζω ότι αποτελούν μέρος μιας δέσμης προτάσεων που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η γνωμοδότησή σα, λοιπόν θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και θα ήθελα ή δυνατόν να μπορέσω κι εγώ να συμβάλλω. Όχι για να σας υποδείξω ότι πρέπει να πείτε εσείς ως Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων, αλλά περισσότερο για να σας πω ότι θα ήταν χρήσιμο όσον αφορά την ίδια τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων σε σχέση με τη δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης, ζητήματα που έχετε ήδη θίξει. Καταρχάς να αφαιρθώ στο ζήτημα του χρονοδιαγράμματος με τον κύριο Μπέγκε, ο οποίο είναι συνεισηγητής και αυτό. Θέλουμε πάντα να έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό μας φέρνει σε τεραχρονισμό με τις πραγματικές ανάγκες. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουμε το δημοψήφισμα στον Ηνωμένο Βασίλειο και όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε μέχρι το τέλος του 2016. Προκειμένου η δική μας συμβολή λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι αποτελεσματική, πιστεύω ότι θα πρέπει πιστά να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα που δεν είναι βέβαια αυτό το οποίο είχαν κατά νου αρχικά οι πέντε πρόεδροι όταν συνέταξαν τη δική τους την έκθεση. Στην περίπτωση αυτή οι πέντε πρόεδροι προέβλεπαν ένα πολύ πιο διαφορετικό χρονοδιάγραμμα το οποίο σχετιζόταν περισσότερο με το πολιτικό θεματολόγιο το εθνικό παρά από τις εξελίξεις που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμείς αν ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα αυτό θα καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ε, την επαύριο του Βρετανικού Δημοψηφίσματος θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τόσο υπόθηκαν σε σχέση με αυτό, απλώς να προσθέσω ότι αν τελικά επικρατήσει το ναι, πράγμα το οποίο είμαστε θεωρώ όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, αν επικρατήσει λοιπόν το ναι στο δημοψήφισμα της Βρετανίας, τότε η ε, συμφωνία αυτή που έχει αυτή τη στιγμή συζητηθεί θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει. Και θα προβλέπετε ότι δεν θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει το δικαίωμα αρνησικυρίας όσον αφορά την ε, ολοκλήρωση της Ευρωζώνης. Τα όσα λέγονται αυτή τη στιγμή θεωρητικά δεν ξέρω τι μορφή θα πάρουν στην πράξη. Θα πρέπει λοιπόν εξ αρχής εμείς να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε το η Βρετανία να ουσιαστικά μάλλον να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που ενδεχομένω να προκύψουν από τη νέα αυτή συμφωνία παρακάμπτοντας το ίδιο το νοσιακό δίκαιο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να παρακάμψουμε την κοινοτική μέθοδο για να προχωρήσουμε όλο και περισσότερο σε μια διακυβερνητική μέθοδο που θα έχει ως αποτέλεσμα τελικά να παρακαμφθεί ακόμα περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει εξ αρχής να ξεκαθαριστεί. Όσον αφορά τώρα την ενσωμάτωση της δημοσιονομικής αυτής ικανότητας της Ευρωζώνης στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, πρέπει εδώ πέρα να είμαστε κάπως δημιουργικοί, ενδεχομένως νομομαθείς να μπορούν να μας βοηθήσουν. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα μέσα, τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη δημοσιονομική ικανότητα και να την εντάξουμε και στον προπολογισμό των γενικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα γίνει με το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, αυτό μου απασχολεί περισσότερο. Πρόκειται όντω για ένα πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο με ανώτατο όριο, χωρί εδώ πέρα να προβλέπεται η δυνατότητα προσαρμογή βάσει των ε, εξελίξεων που ενδεχομένω θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο άμεσο διάστημα. Πράγμα το οποίο αναγκαζόμαστε να κάνουμε πολύ συχνά. Δεν ξέρω λοιπόν αν εδώ πέρα θα προκύψουν κάποια προβλήματα όταν θα πρέπει να αυξήσουμε το ανώτατο αυτό όριο για να ανταποκριθούμε σε κλειδονισμούς που μπορεί να προκύψουν στα πλαίσια του κοινοτικού προπολογισμού. Αναφερθήκατε επίσης στο EFSM. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει και πάλι εδώ πέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστικής Σταθερότητας και τι μπορούμε να κάνουμε και με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, τον ESM στην έκθεση των πέντε προέδρων προβλέπεται σε ένα μεταγενέστερο στάδιο να δούμε πώς θα καταφέρουμε να ενσωματώσουμε στη νέα αυτή δημοσιονομική ικανότητα στον προπολογισμό τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ESM. Αυτό ήταν μια αρχική πρόθεση η οποία είχε εκφραστεί και στην έκθεση των πέντε προέδρων και πρέπει πιο έμπρακτα τώρα να ασχοληθούμε και με το ζήτημα αυτό. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σα δώσω περισσότερε λεπτομέρειε, απλώ σα καλώ να βαθύνετε και περισσότερο. Τρει ακόμα παρατηρήσει. Πρώτον, όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια λέτε στο σχέδιο γνωμοδότησής σας, στο προσωρινό αυτό σχέδιο γνωμοδότησης, ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της επικορικότητας. Πολύ ωραία. Αν όμως αρχίσουμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε όλο και περισσότερο για αυτή τη δημοσιονομική ικανότητα και τελικά τη θεσπίσουμε, δεν μπορούμε να μείνουμε και να αρκεστούμε στο εφιστάμενο πλαίσιο. Κάτι περαιτέρω, κάτι παραπάνω θα πρέπει να προβλέψουμε και εδώ θα πρέπει να είμαστε δημιουργικοί, αλλά δεν μπορούμε να παραμείνουμε στο εφιστάμενο πλαίσιο. Αναφερθήκατε επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ με τα όσα είπατε. Δεν λέω ότι θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν προτείνεται άλλωστε κάτι τέτοιο. Να δούμε όμως τι μέσα εποπτείας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να εμπνευστούμε από τα μέσα εποπτείας τα οποία προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε και για την Ευρωζώνη. Αυτή τη στιγμή η διάκριση που γίνεται μεταξύ χωρών εντό και εκτό Ευρωζώνη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όσον αφορά τώρα την διοικητική δομή, την εκτελεστική δομή αυτή τη δημοσιονομική ικανότητα Ευρωζώνη, ανέκαθεν λέγαμε ότι θέλαμε έναν Υπουργό Οικονομικών, αυτό έλεγα εγώ πάντα, ένα Υπουργείο Οικονομικών της Ευρωζώνης και ότι ε, οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να υπάγονται στον Αντιπρόεδρο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιος για το ευρώ. Ένα λεπτάκι ακόμα μπορείτε να μου δώσετε και ολοκληρώνω. Έχω την εντύπωση ότι κάποιοι θεωρούν ότι μακρηγόρησε. Ολοκληρώντας λοιπόν, στο ενδιάμεσο αυτό διάστημα στο οποίο μπαίνουμε σιγά σιγά, αν θέλουμε πραγματικά να διατηρήσουμε ένα υψηλό βαθμό φιλοδοξίας και να κάνουμε και συγκεκριμένε προτάσεις οι οποίες όντως θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από το Συμβούλιο, διερωτάμε λοιπόν αν η διαχείριση ενός προπολογισμού της Ευρωζώνης δεν θα πρέπει ουσιαστικά να συνάδει να εμπνευστεί από το σύστημα διαχείρισης, τη διάρθρωση διαχείρισης της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ξέρετε ότι έχουμε τον πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας, ένα διοικητικό συμβούλιο και ένα διαχειριστικό συμβούλιο. Δεν λέω ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε το σύστημα αυτό ακριβώς έτσι στα πλαίσια του α, κοινοτικού πλαισίου. Από την άλλη όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες συναφείς προτάσεις, ανάλογες προτάσεις, προκειμένου να καταλήξουμε πραγματικά στην ευκταία διάρθρωση που θα θέλαμε να έχουμε για αυτή τη δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης, η οποία να μπορεί όμως να λειτουργήσει και στην πράξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου δώσατε, Προτιμώ να καταφέρω και εγώ να εκφράσω την άποψή μου στα πλαίσια της ζήτησης αυτής. Μας έβαιναν δύο ακόμη μιλητές, ο Έλμαρ Μπρόκ και ο Πέντρο Περέρα. Στο τέλος θα δευτερολογήσει ο εισηγητής μας. Συμφωνούμε σκέφτομαι λοιπόν πως είναι δυνατόν να τα καταφέρουμε αυτά, αλλά επιτρέψτε μου κάποιες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι όπως ο συνάδελφος Ρανζέλ έχει αναλάβει αυτή την έκθεση, είναι μια σημαντική έκθεση και θα τα καταφέρει καλά. Θέλω να ευχαριστήσω για την προσπάθειά του. Θέλω όμως να τονίσω ότι η δομή, η θεσμική δομή θα έχει επιπτώσεις και δεν μπορεί να επαφεθεί μόνο στον πλούτο επιχειρημάτων και ιδεών των μελών της ΕΚΟΝ διότι ίσως αυτό περιορίζει τα πράγματα σε σχέση με ένα ευρύτερο πλαίσιο και νομίζω ότι και εμείς ε, εδώ τώρα δεν θα ασχοληθούμε με το ποιος, ε, με το τι ακριβώς θα γίνει με τα χρήματα αυτά, πράγμα που είναι δική τους αρμοδιότητα. Το θέμα με το Κοινοβούλιο είναι σημαντικό. Έχουμε προτάσεις ε, από πλευράς του εγγράφου των πέντε προέδρων. Έχουν γίνει προτάσεις και σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο και με άλλες αφορμές. Αυτά τα οποία εκφράστηκαν, ότι δηλαδή ο συνάδελφος ε, δεν είναι εδώ, ότι πρέπει να προσέξουμε σαφέστερα να μην υπάρξει σύγχυση αρμοδιοτήτων, ενίσχυση των, ε, εθνικών κοινοβουλίων μέσα στο πλαίσιο της ελεγκτικής τους δραστηριότητας, εκεί όπου έχουν αρμοδιότητες κοινοβουλευτικά, στο εθνικό πλαίσιο και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο οι ελεγκτικές αρμοδιότητες να είναι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μην συγχαίουμε δηλαδή τα πράγματα αυτά. Στον ρόλο του Ευρωπαϊκού λοιπόν Κοινοβουλίου πρέπει να είναι σαφές ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει αυτό να αποτελέσει τμήμα του γενικού προϋπολογισμού. Ο ειδικό προϋπολογισμός δηλαδή για τα δημοσιονομικά, για την δημοσιονομική ικανότητα και όταν θέλουμε λοιπόν να υπάρξει η ε, ρύθμιση αυτή δεν μπορούμε ξεχωριστά να καταλήξουμε σε μια ξεχωριστή έκτακτη λύση όπως με το Ταμείο Ανάπτυξης ε, που ε, επί χρόνια γίνεται η προσπάθεια να ενταχθεί στο σωστό πλαίσιο. Πρέπει να προσέξουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο τεχνικά μπορεί να υπάρξει μια τέτοια δυνατότητα το earmarking, ο προκαθορισμός δηλαδή κονδυλίων ε, μπορεί να ε, λειτουργήσει κανονικά ως ήθιστε και έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν να ενταχθεί αυτό στο γενικό προϋπολισμό υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υποβάλλω μια πρόταση να σκεφτούμε και να δούμε αν αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ευρωχώρες, τις ευρωζώνης δηλαδή τις χώρες ή και για ειδικές, ε, ειδικά για χώρες που προετοιμάζονται εντονώς για να ενταχθούν στην Ευρωζώνη. Και μπορεί αυτό να είναι ένα κίνητρο για αυτές τις χώρες, ε, για μια μεταβατική περίοδο για αυτές προς το, προς το ευρώ, δηλαδή για κάποιες χώρες που δεν είναι χώρες της Ευρωζώνης σήμερα και θα μπορούσαν ε, να ε, δρομολογήσουν την ένταξή τους στην Ευρωζώνη, ώστε να μπορέσουν έτσι να έχουν μια, ένα ενθαρρυντικό κίνητρο να δράσουν. Αλλά θα πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι όπως πολλές φορές υπό μεγάλη πίεση επιτυχάνεται, αυτό να μην αποτελέσει διαφοροποίηση θεσμική μεταξύ χωρών της Ευρωζώνης και μη χωρών της Ευρωζώνης. Και το έγγραφο για, την, για το Brexit, για την ε, ε, αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται ότι δεν πρέπει να γίνεται με ε, διαφοροποίηση μεταξύ χωρών Ευρωζώνης ε, και μη χωρών Ευρωζώνης ε, αλλά χωρών που θα ενταχθούν στην Ευρωζώνη και χωρών που βρίσκονται στην Ευρωζώνη σήμερα. Δηλαδή ότι η υλοποίηση των υποχρεώσεων από αυτές τις χώρες είναι αεπιτακτική ανάγκη και αναφέρεται και στο έγγραφο Brexit ότι η Μεγάλη Βρετανία ως μέρος της ε, ενιαίας εσωτερικής αγοράς θα έχει δυνατότητες ενημέρωσης και πληροφόρησης και θα έχει και το, τη δυνατότητα συζήτησης αυτών των θεμάτων στο Συμβούλιο ώστε να υπάρχει ενημέρωση για τα μειονεκ... ώστε να αποφύγουν μειονεκτήματα ε, για... όσον αφορά την ενιαία εσωτερική αγορά για λογαριασμό τους. Όμως δεν θα έχουν δικαίωμα αρνησή κυρίας, δεν θα έχουν δικαίωμα βέτο και σε σχέση με την πρόταση που θα υποβάλλεται στο Συμβούλιο Υπουργών πλειοψηφικά θα λαμβάνεται απόφαση επιθεμάτων που αφορούν τη δική τους δικαιοδοσία. Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν κάτι αντίστοιχο να συμβεί και πρέπει να επιμείνουμε και να εμείνουμε ότι ρητά αυτό αφορά το, την ικανότητα ανάπτυξης της Ευρωζώνης περαιτέρω. Συμφωνία με τους Βρετανούς αναφέρεται ρητά ότι οι Βρετανοί δέχονται ότι μπορεί να εμβαθυνθεί η Ευρωζώνη περαιτέρω και δεν θα έχουν ένσταση ή κάποια αντίρρηση. Πρέπει λοιπόν επ' αυτού να βασιστούμε και έτσι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε Εντάξει, δεν θέλουν σε κάτι να συμμετάσχουν πολύ καλά, αλλά συζητάμε και στη Γερμανία για παράδειγμα για ειδικέ τέτοιες ε, ε, δυνατότητες και πιστεύω ότι πρέπει να θεωρήσουμε σημαντικό το θέμα της μετεξέλιξης μετεξέλιξης των θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων και έτσι πρέπει να διασφαλιστεί ότι το Single Framework Unit θα μπορέσει να προ, προαχθεί. Το ερμηνεύω ότι δηλαδή δεν θα, μπορέσουν, δεν θα μπορέσουν άλλοι να εμπλέκονται και ε, όσον αφορά τους υπουργούς οικονομικών και εδώ πρέπει να επαναλάβουμε το αίτημα που και οι Μερθέντες και εγώ έχουμε διατυπώσει την έκθεσή μας και που ανήκει σε αυτό το πλαίσιο, ότι δηλαδή ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για οικονομικά και νομισματικά θέματα, θα είναι ο επικεφαλής της Ευρωζώνης. Το επιτρέπει αυτό η συνθήκη και μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Και έτσι με ένα μπάρο δυο τριγώνια πολλά προβλήματα θα διευθετήσουμε αντί από πλευράς ε, νέων Υπουργών Οικονομικών, νέος Πρόεδρος να προσδιοριστεί Νομίζω λοιπόν αυτό θα δημιουργούσε κάποιο πρόβλημα, χάος στη διοίκηση ε, και διευθέτηση αυτών των θεμάτων. Μπορούμε λοιπόν εδώ να διασυνδέσουμε το θέμα με αυτόν τον τρόπο προτείνοντας ε, την άλλη εναλλακτική λύση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ίσως αυτό μπορεί να μην είναι η δική τους πρώτη προτεραιότητα, αλλά αυτό πρέπει να προταθεί σε σχέση με την ε, Ευρωομάδα, ώστε να διευθετηθούν τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Ελμάρο Πέντρο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον Πάολο Ραντζέλ. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι το θέμα είναι και σημαντικό αλλά και δύσκολο. Πολλό δε μάλλον στο στάδιο που βρισκόμαστε. Και εν ώψη του δημοψηφίσματος ε, της Μεγάλης Βρετανίας. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε τι προσθέμενη αξία μπορούμε να δώσουμε εμείς στην πρόταση αυτή ως Επιτροπή Στεγματικών Υποθέσεων. Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην συζήτηση, στον εμπλουτισμό της, με τις συγκεκριμένες προτάσεις. Και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι σε αυτή τη φάση είναι πολύ δύσκολο να είμαστε πολύ πλήρεις ε, και συγκεκριμένοι με τις προτάσεις μας. Έχουμε εδώ πολύ σημαντικές πολιτικές δηλώσεις που λένε ότι χρειαζόμαστε δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης και θα πρέπει να τη δημιουργήσουμε, αυτή η ικανότητα η δημοσιονομική τη Ευρωζώνη θα πρέπει να αποτελεί τμήμα του γενικού προπολογισμού να λαμβάνεται υπόψη η νομοποίησή τη και να εξασφαλίσουμε την ανάμειξη των εθνικών κοινοβουλίων. Τώρα για τα συγκεκριμένα θέματα λαμβάνουμε υπόψη τις διαφορετικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί και αναγνωρίζουμε ότι ακόμη και κράτη εκτό τη Ευρωζώνη θα πρέπει να εμπλακούν στη διαδικασία, αλλά με διαφορετικό τρόπο από ότι τα κράτη-μέλη τη Ευρωζώνη. Αλλά αυτή τη συζήτηση θα τη συνεχίσουμε και στο μέλλον. Αυτές οι πολιτικές διακηρύξεις νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό θέμα και η πιο σημαντική συμβολή της Επιτροπής μας σε αυτή τη φάση. Στο μέλλον θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε και εναλλακτικέ προτάσεις και κυρίως να αναλύσουμε τις θεσμικές συνέπειες των επιμέρους ε, προτάσεων. Αυτή δεν είναι η προστιθέμενη αξία και η δική μας προσφορά και συμβολή στη συζήτηση. το πώς θα εμπλέκονται οι χώρες εκτός Ευρωζώνης στην όλη διαδικασία θα το δούμε στο μέλλον. Επίσης, πώς θα διασφαλίσουμε την ένταξη κάποιων κονδυλίων ή ταμείων, όπως το ΕΦΣΥ και το παιδικό σχέδιο του Ιουνκέρ στον προϋπολογισμό. Όλα αυτά τα θέματα είναι ανοιχτά προς συζήτηση. Πάντως, το εναρκτήριο λάκτισμα που δόθηκε είναι πολύ θετικό. Σας ευχαριστώ. Ο Πάολο Ραζέλ τώρα, θέλεις, θέλεις να δευτερολογείς. Τρία λεπτά έχεις μόνο όμως. Καλώς, ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση της ε, Mercedes Μπρέσο και της Σιλβί Γκουλάρ. Ότι η γνωμοδότησή μας θα πρέπει να είναι φιλόδοξη. Βέβαια, όχι επί παντός επιστητού, αλλά να καλύπτει ένα φάσμα απόψεων που θα αντανακλάται και στην έκθεση εικόν. Συμφωνώ λοιπόν με αυτή την προσέγγιση. Εμένα δεν απασχολεί τόσο η έκβαση του δημοψηφίσματος και το Brexit, γιατί ως προς αυτό θα έχουμε πολλές συνέπειες, ακόμη και σε περίπτωση αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας. Κύριε Μέσερ Σμιτ, θα ήθελα να σας πω ότι στο σημείο 5 προβλέπουμε καθορισμού νέων κατηγοριών ιδίων πόρων, ακόμη και προέρχονται μόνο από ένα κράτος μέλος. Εννοείται ότι για, την, για τον προπολογισμό της Ευρωζώνης θα λαμβάνονται συνεισφορές μόνο από χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό είναι λογική απόρρεια. Και έτσι ξεπερνάμε και το, το βρετανικό ζήτημα. Επίσης, η ιδέα ότι θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι θα εξαρτηθεί και από τις λειτουργίες που θα αναγνωρίσει η ΕΚΟΝ στη δημοσιονομική ικανότητα. Η συγκεκριά κυρία Περβάνς Περές πέφτει έκκληση και στο ρεαλισμό μας. Συμφωνώ, γιατί μερικές φορές ε, αν ε, δεν είμαστε ρεαλιστέ, δεν έχουμε πιθανότητε να ευοδοθούν. Θα πρέπει να συνδυάσουμε ρεαλισμό και φιλοδοξία για να μην έχουμε ένα απλό ευχολόγιο. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των φιλοδοξιών μα και του δυνατό εφικτού και του ρεαλισμού που μπορεί να γίνει δεκτό και από άλλου. Έτσι έχουμε και περισσότερε πιθανότητε να γίνει δεκτή η γνωμοδότησή μα. Τώρα, για το αν θα πρέπει να πρόκειται για Ευρωπαίο Υπουργό ε, Οικονομικών ή Ευρωπαϊκό Διοικητικό Συμβούλιο, ένας υπουργό ε, οικονομικό θα πρέπει να είναι μέλος, ε, αν θα πρέπει να είναι μέλος Επιτροπής. Αυτό σε μεταγενέστερο επίπεδο όμως ε, θα τα, θα τα δούμε. Και αυτό και άλλα θέματα. Ίσως μόνο σε, στη φάση των τροπολογιών. Γιατί αυτή τη στιγμή λόγω του περιορισμού των χαρακτήρων δεν μπορούμε να καλύψουμε όλη την περιπλοκότητα του θέματος. Το είπε και η Μερσέδες. Κάτι που επίσης θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι καλό θα είναι να έχουμε κάποια σύμνοια με άλλες εκθέσεις, ιδιαίτερα την έκθεση Μπρέσο Μπρόκ. Να έχουμε κάποια εναρμόνιση, ευθυγράμμιση, αν προλάβουμε. Μάλλον προλαβαίνουμε, χρόνο έχουμε. Τώρα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, που δεν ήθελα να πω ότι θα πρέπει να αναμειχθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Απλώς είπα ότι μπορούμε να εμπνευστούμε από ένα μοντέλο διαφοροποίησης ε, κατά το πρότυπο της ΕΚΤ. Μια διαφοροποιημένη λύση δηλαδή μεταξύ χωρών Ευρωζώνης και ε, χωρών εκτός Ευρωζώνης. Σε περίπτωση που τα μέλη εκτός Ευρωζώνης θέλουν να συμμετέχουν. Αυτή είναι η ιδέα. Και συμφωνώ με τον κύριο Μέσσερ Σμιτ να διαφυλάξουμε οπωσδήποτε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κάτι τέτοιο όμως δεν αποκλείει να έχουμε τακτικές επαφές με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΤ ε, για να εξασφαλίσουμε ένα είδος λογοδοσίας. Κάτι που δεν έχει όμως σχέση, δεν επεμβαίνει σε καμία περίπτωση με την ε, ε, ανεξαρτησία της Στις 28 θα συνδεθώ με τα μέλη της ΕΚΟΝ και θα σας υποβάλω την οριστική εκδοχή του σχεδίου και θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε και να καταθέσετε και τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι στις 5 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσει η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Εμείς θα πρέπει να ψηφίσουμε στις 12 Ιουλίου τη δική μας γνωμοδότηση εδώ. Αν όμως ε, καθυστερήσει, αναβληθεί η ψηφοφορία στην Επιτροπή Budget και ΕΚΟΝ, μπορούμε και εμείς να το αναβάλουμε, αλλά πρέπει να περιμένουμε. Ναι, για μένα είναι δύσκολο, γιατί δεν θα είμαι εδώ 12 Ιουλίου. Θα είμαι στη Washington. Βλέποντας και κάνοντας. Δεν είμαι σίγουρος πάντως. Καλά, θα το δούμε. Πάντως με βάση το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα, εμείς θα ψηφίσουμε 12 Ιουλίου. Οπότε η εξέταση των τροπολογιών μπορεί να γίνει στις 15 Ιουνίου. Είπατε ότι το Μάιο θα αποσιάζεται, οπότε δεν θα γίνουν άλλες συζητήσεις. Θα έχουμε απλώς εξέταση τροπολογιών. Και έχουμε και μακρά διορία για την υποβολή των τροπολογιών. Να έχουμε και τη συμβαστική με πρόταση του ΕΛΚ. Οπότε, 7 Ιουνίου το μεσημέρι λίγη προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. 7 Ιουνίου. Μέχρι τότε μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες. Και 15 Ιουνίου θα γίνει εξέταση των τροπολογιών προκειμένου να ψηφίσουμε τον Ιούλιο, αν δεν υπάρξουν αλλαγέ. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, έκθεση, γνωμοδότηση μάλλον του Πέντρου Σίλβα Περέιρα για τη μετεκλογική αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, θα τη δούμε το απόγευμα, θα είναι το πρώτο σημείο αμέσω μετά τις ψηφοφορίες. Έκθεση του κυρίου Σίλβα Περέιρα. Διακοπή μέχρι το απόγευμα.